tanta gente. Buenas tardes. Γεια σας. Ας ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δυστυχώς ε, έχουμε πολύ λίγες παρουσίες από πλευράς ευρωβουλευτών. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι όπως θα είδατε τα σημεία 5 και 6 μερίσιας διάταξης για το γάδο ε, μετατέθηκαν για αύριο στις 19 του μηνός γιατί η κυρία Ντότς δεν ήταν εύκαιρη σήμερα. Θα αντικατασταθούν από το σημείο 17 έκθεση Ρωμέβα. Ο κύριος Ρωμέβα συμφωνεί πήραμε τη γνώμη του. Οπότε αυτή είναι η πρόταση που σας κάνω, αν συμφωνείτε. Είχα πει και παλιότερα ότι, και το λέω ξανά, εδώ όχι μόνο στους συντονιστές για να είναι παρόντες συνάδελφοι, είναι η τελευταία φορά που αλλάζουμε την Μέση διάταξη χωρίς σοβαρό λόγο. Γιατί τελευταία ο καθένα όπω τον βολεύει ζητά τελευταία στιγμή αλλαγή τη ημέρησια διάταξη. Αυτό ε, είναι σε βάρο της ε, επιτροπή ε, των άλλων Ευρωβουλευτών και των τεχνικών μας υπηρεσιών. Οφελεί μόνο αυτόν που το ζητάει. Συνεπώς το λέω ξεκάθαρα. Δεν πρόκειται να δεχτώ καμία άλλη αλλαγή τη διάταξης παρά μόνο για έκτακτες περιστάσεις και έκτακτους λόγους. Τώρα, πριν δημοσιευθεί η Μέση διάταξη, θα προσπαθήσει η γραμματεία, θα προσπαθεί η γραμματεία να είναι σε επαφή με όλους προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι ανάγκες. Όμως δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε κάθε φορά ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης την αλλαγή της, την τροποποίησή της. Τελευταία φορά. Αλλαγές θα γίνονται μόνο κατ' εξαίρεση. Νομίζω ότι με αυτόν τον ε, τρόπο θα δώσουμε και περισσότερη αξία στη δουλειά μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι εδώ και τις δύο μέρες. Όχι μόνο όταν τους ενδιαφέρει ένα θέμα ή όταν είναι το θέμα τους. Λοιπόν, δεχόμαστε την τροποποίηση μέσης διάταξης. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι σε σχέση με την έγκριση των πρακτικών της 21 η και 22ης Ιανουαρίου, οι μεταφράσεις δεν είναι έτοιμες, συνεπώς αναβάλλεται αυτή η έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασής μας. Θα γίνει το Μάρτι. Ενημερωτικά απλώς Πρόεδρου. Να σας πω το εξή που το ξέρετε ήδη σίγουρα. Όμως καλό είναι να το ξαναθυμηθούμε. Σα το είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, όχι, σε μια συνεδρίαση συντονιστών το είπα. Πρόταση ψηφίσματος για την ε, μερών της, ε, ε συνάντηση των μερών της σύμβασης ΣΥΤΕΣ. Το υιοθετήσαμε στην προηγούμενη Ολομέλεια. Έχει κάποια ζητήματα, κάποιες πτυχές οι οποίε έρχονται σε πλήρη αντίθεση, με αυτά που έχουμε πει στο παρελθόν. Και ε, ζητήσαμε την παρουσία του Επιτρόπου Περιβάλλοντος εδώ και κάναμε και μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια. Σας το θυμίζω. Προκειμένου ενδεχομένω να λάβουμε κάποια πρωτοβουλία, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το ξαναδούμε. Αύριο. Το σημείο 9 της ημερησίας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο, θα λάβει χώρα και κλεισμένων των θυρών. Ε, δεν το είχαμε ξεκαθαρίσει προ... παλιότερα, το ξεκαθαρίσαμε τώρα, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Για να συζητήσουμε όλα τα ενδιαφέροντα θέματα με άνεση. Υπάρχουν ερωτήσεις, απορίες. Όχι. Περνάμε στο σημείο 4. Α, κυρία Φράγα. Σε σχέση με το θέμα της ΣΥΤΕΣ. Εγκρίθηκε τις προάλλες αυτό το θέμα που το οποίο εμεί διαφωνούσαμε πάντοτε και που είχε σχέση με τις πιστοποίησεις. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, όταν συζητάει θέματα ΣΥΤΕΣ πιστεύω και όταν αυτά τα θέματα έχουν σχέση με την Αλία ε, θα πρέπει να είναι σε επαφή μαζί μας. Ε, έκανε μια πρόταση που υποστήριζε το έγγραφο μέσω του οποίου γίνεται πιο ευέλικτη η χορήγηση πιστοποιήσεων. Εμείς διαφωνούμε όμως με αυτό. Ε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος ξέρει πολλά για την αλία, αλλά όχι και τόσο όσο εμείς. Οπότε όταν εκδίδονται ψηφίσματα ΣΥΤΕΣ που περιλαμβάνουν ζητήματα αλίας, θα πρέπει να συντονιζόμαστε, γιατί δεν είναι δυνατόν εμείς εδώ πέρα να λέμε στους επιτρόπους δεν γίνεται το ένα δίνει το άλλο και μετά η Επιτροπή Περιβάλλοντος να κάνει τα δικά της. Και ε, έκανε τα δικά τη γιατί δεν γνωρίζει το θέμα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να του εξηγήσουμε. Αν του είχαμε εξηγήσει, σίγουρα θα μα είχαν πιστέψει, θα είχαν πιστεί. Δεν είναι δυνατόν να ε, υποστηρίζει μια ε, πρόταση η οποία ε, είναι εναντίον της πολιτικής μας για την καταπολέμηση τη παράνομη και άναρχης Συνεπώ, Συνεπώς, προσοχή για αυτά τα θέματα, ιδιαίτερως για ζητήματα ΣΥΤΕΣ, που είναι η επικεφαλής η ομάδα περιβάλλοντος και ποτέ δεν ζητάει τη γνώμη μας. Θέματα τέτοιου τύπου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ωραία. Οπότε, δύο θέματα. Ε, να είμαστε σε επαφή με την γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και εγώ θα μιλήσω με τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής προκειμένου να, η σχέση μας να είναι πιο τακτική ε, έτσι ώστε να συντονιζόμαστε. Χωρίς να περιορίζεται βέβαια η ελευθερία κατέρωθεν. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ έχουμε δύο από τους συντονιστές της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος και δεν νομίζω ότι αυτοί δεν θέλουν να συνεργάζονται μαζί μας. Αυτό θα ήταν ε, ενάντια στα συμφέροντά μας. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που σαφώς πρέπει να διαφυλάξουμε είναι η επικοινωνία. Σημείο 4. Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας. Εισηγητής ο κ. Καντέκ. Ε, προθεσμία τρόπο η αποβολή του έχει λήξει. Υποβλήθηκαν 2.445 τροπολογίες. Ε, η Επιτροπή Ντέβερ έχει, Έμπλ και λοιπά ε, και Έμβη υπέβαλαν επίσης τροπολογίες. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν αυτές τις ε, ε, τροπολογίες. Θα δώσω το λόγο κατευθείαν στον εισηγητή μας, τον κύριο Καντέκ. Και βέβαια στους υπόλοιπους συναδέλφους. Euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε, 2.445 τροπολογίες. Ορίστε, 400 τροπολογίες των επιτροπών που ήταν υπεύθυνε για γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ για όλη την εργασία που επιτελέσατε για να αποκτήσουμε αυτό το τόσο εκτενή φάκελο. Και καταλαβαίνετε τι δουλειά σημαίνει αυτό και για τον εισηγητή και για τους και εισηγητές. Σας ευχαριστώ ούτως ή άλλως, διότι αυτό σημαίνει ότι σας αφορά πάρα πολύ το θέμα αυτό. Δεν είχα και καμία αμφιβολία βεβαίως. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρώτη μου παρατήρηση θα είναι η πρωτη μου παρατηρηση ειναι η εξη Εφ' εξής, η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο Θάλασσας και Αλληγίας θα γίνει μετά την ε, ψήφιση του βασικού κανονισμού, όπως είχαμε πει στην τελευταία Ολομέλεια ψηφίστηκε στο Στρασβούργο Και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι με ικανοποίηση είδα ότι δεν υιοθετήθηκε η αρχή των ε, θέσεων κάτ εξουσιοδότηση που παρέχονται σε άλλους για να αλλιεύουν. Επίσης, ξέρουμε ότι έγινε ε, δεκτή, δεκτό το θέμα της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Όπως ξέρετε, οι περισσότεροι ευρωβουλευτές θέλησαν αυτή την υποχρέωση εκφόρτωσης να την καταστήσουν υποχρεωτική, το λαμβάνουμε υπόψη και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να το εντάξουμε στα πλαίσια του ΕΤΘΑ. Έγινε μια πρώτη συνάντηση των σχεδόν συντονιστών για να μπορέσουμε να ενθεσπίσουμε τη μέθοδο εργασίας την οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Συμφωνήσαμε για κάποιες αρχές που θα μας επιτρέψουν, ελπίζω, να λειτουργήσουμε με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τις καλύτερες δυνατές συνενετικές ίσεις. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε μόνο εγώ και οι σκιώδεις ηγητές, οποιοδήποτε βουλευτής μπορεί να συζητήσει την οποιαδήποτε τροπολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να πει ποια είναι η άποψή του. Πιστεύω λοιπόν ότι στα σχέδια στο σχέδιο της έκθεσης που σας ε, υπέβαλα βάσει της πρότασης Επιτροπής θέλησα να επικεντρωθώ σε δύο προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα η διάρκεια. Με την ευρία της έννοια, συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή η επιθυμία μας είναι να μπορέσει να είναι βιώσιμη στο χρόνο η ευρωπαϊκή αλία σε όλους τους τομείς. Περιβαλλοντικό, ε, κοινωνικό και οικονομικό βεβαίως άρα και ανταγωνίσιμη ανταγωνιστική. Το πρώτο σημείο λοιπόν, η διάρκεια στο χρόνο, στο εγγραφό μου, επιμένω ότι είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητες ε, επενδύσεις όσον αφορά τα διάφορα λιευτικά εργασία, η υποχρέωση ε, εκφόρτωσης ε, ε, με τρόπο που να αποφεύγονται οι απορρίψεις, δηλαδή να προσπαθήσουμε να έχουμε με επιλεγμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε λιγότερες απορρίψεις. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι πρωταρχική σημασία. Πρώτη παρατηρήση μου. Δεύτερη, να διευκολυνθεί η υιοθέτηση σχεδίων διαχείρισης. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο και κανένας δεν έχει μεγάλες αντιρρήσεις επί του θέματος αυτού. Επίσης, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει τις προσωρινές παύσεις και μετά θα δούμε βάση ποιων κριτηρίων και όρων. Όσον αφορά λοιπόν τη διάρκεια στον χρόνο αυτής της δραστηριότητας ελληνικής για την Ευρώπη, θα ήθελα να είμαστε απολύτως σαφείς σε κάποια πράγματα. Είμαι εντελώς αντίθετο σε οποιαδήποτε επένδυση που θα αυξήσει την ε, ε, αλληλευτική ικανότητα. Μην ε, νομίσει κανείς ότι θέλω κάτι τέτοιο, δεν το είπα ποτέ. Σήμερα πιστεύω ότι η ελευθερική ικανότητα, η ικανότητα της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πάρα πολύ καλά καθορισμένη, σε γενικές ε, γραμμές δεν προβλέπει πλεόνασμα αυτής της ικανότητας. Θα ήθελα επίσης να μπορέσουμε κάποια κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας να τα διαθέσουμε για να γίνει σεβαστό αυτό από τα κρατημέλη. Πιστεύω ότι θα πρέπει εξάντε εκ των προτέρων, όπως έγινε στην Επιτροπή ΔΕΒΗ για τα άλλα κοινοτικά κονδύλια, να το θέσουμε ως προϋπόθεση. Και προσδίδω ιδιαίτερη σημασία, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι με το οποίο συμφωνείτε όλοι σας, στους ελέγχους και στην συλλογή δεδομένων, διότι πιστεύω ότι είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει την διάρκεια στον χρόνο όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Αλίας. Αρνούμε αυτό το χρηματοδοτικό μέσο να χρησιμοποιηθεί για την ανασυγκρότηση των αλλιέων υπό την ετοιμολογική έννοια. Απ' την άλλη, απ την άλλη όμως να γίνει ένα μέσον ε, για να μπορέσουν να ασκήσουν κάποιες συμπληρωματικές δραστηριότητες οι αλληλείς είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνο. Η ανασυγκρότηση όμως είναι πάρα πολύ σπαστικός όρος και μπορεί να φοβήσει κάποιους, διότι ίσως κάποιοι πιστεύουν ότι θέλουμε τους αλληλείς να τους κάνουμε να αλλάξουν επάγγελμα, να ακολουθήσουν ένα άλλο επάγγελμα. Γι' αυτό είναι μακρά εμού στην πρόταση αυτή. Η συμπληρωματικότητα, η διαφοροποίηση είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ, αλλά τίποτα περισσότερο. Επίσης, θα ήθελα να θεσπίσουμε μία βοήθεια για την εγκατάσταση των νέων αλλιέων για αυτό το επάγγελμα. Το ωραίο, αλλά σκληρό επάγγελμα. Και βεβαίως, συγχρόνως, να γίνουν επενδύσεις και σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης. Μου φαίνεται ότι αυτό είναι απαραίτητο. Και βεβαίως, το τελευταίο σημείο, το οποίο είναι ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένω θα υπάρξουν αντιθέσεις, το είδαμε αυτό να αντικατοπτρίζει σε πολλές τροπολογίες, είναι το θέμα των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου της Ευρώπης, που υπενθυμίζω, για όσους δεν το έχουν ακούσει εδώ και 3,5 χρόνια, σχεδόν 4, σήμερα κατά μέσον όρο έχει ηλικία 27, 28 χρόνια θα έλεγα. Απ' την άλλη, θα ήθελα να πω ότι και ακόμη μία φορά με τις επιφυλάξεις τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Και πιο σημαντική είναι ανανέωση του αλευτικού στόλου για, τους, για δεδομένου ότι γυράσκει, αλλά χωρίς να αυξηθεί η αλευτική ικανότητα του αλευτικού στόλου της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα σλόγγαν που το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Το επαναλαμβάνω. Και όπως έλεγα, αν δεν έχουμε ψάρια, δεν θα έχουμε κι αλλιείς. Εδώ λέγω, θα πρέπει να αλλιεύουμε καλύτερα και όχι περισσότερο. Αυτή λοιπόν είναι η φιλοσοφία την οποία ακολούθησα στο έγγραφό μου. Πολύ καλά δουλέψατε με τις 2.245 τροπολογίες, διότι είναι μέρος των κανόνων του παιχνιδιού. Εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με τους συναδέλφους, τους και όλους συζητητές, ως για να επιτύχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συμβαστικών λύσεων. Δεν είναι απλά τα πράγματα, το είδαμε και στον ε, αρχικό κανονισμό αυτό, αλλά πιστεύω ότι σε πολλά σημεία θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνίες, σε σημεία σύγκλησης, διότι πιστεύω ότι όλοι, και το ελπίζω τουλάχιστον, εμείς εδώ αυτό το οποίο θέλουμε κυρίως είναι να επιβιώσει η ευρωπαϊκή αλία, η δραστηριότητά της, αυτό επιθυμώ και εγώ, με κάποιες ρυθμίσεις, με κάποιες αλλαγές, όπως είδαμε και στο βασικό κανονισμό, αλλά η βούληση αυτή ούτως ή άλλως πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο συμμερίζεται η πλειοψηφία μεταξύ ημών. Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, κάνουμε ανταλλαγή απόψεων φαντάζομαι και δεν θα αρχίσουμε να εξετάζουμε επιμέρους κάθε μία από όλες τις τροπολογίες που έχουν κατευθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεσή σας, είμαι εδώ για να σας ακούσω και θα αρχίσουμε από μεθαύριο. Η πρώτη συνεδρία με τους χιώδης θα λάβει χώρα μεθαύριο και θα εργαστούμε στις τρεις πρώτες ομάδες τροπολογιών. Υπάρχουν ήδη προτάσεις για συμβαστικές τροπολογίες και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα σημεία. Αυτά ήθελα να πω. Είμαι στη διάθεσή σας, είμαι ως εισηγητής στη διάθεσή σας και στην υπηρεσία σας. Γι' αυτό έχει οριστεί ο εισηγητή. για να είναι στην υπηρεσία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Η κυρία Φράγκα, η κυρία Πατράων και άλλοι συναδελφοί ζήτησαν το λόγο. Bien, tenemos 12 peticiones de... 12 συνάδελφοι ζητούν το λόγο. Πολύ ενεργητικού σας βλέπω. 13, 14. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βολευτούμε με το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Σε πάση περιπτώσει, έχουμε χρόνο σήμερα σήμερα το απόγευμα, εφόσον άλλαξαν κάποια θέματα στη μέρη διάταξη, έχουμε χρόνο. Θα προσπαθήσουμε ούτω ή άλλω να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Δύο-τρία λεπτά, όχι περισσότερα, ο κάθε συνάδελφο. Διαφορετικά δεν θα έχουμε χρόνο για να τελειώσουμε τα σημερινά θέματα. Ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, όσον αφορά τις δικές μου τις ε, τροπολογίες, θα ήθελα να φερθώ στο σχέδιο του κανονισμού και όχι στα εδάφια. Θα ε, εστιάσω την προσοχή μου σε τρεις τροπολογίες που τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Καταρχήν, η 484-32. Έκτο θέμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ε, αλία εσωτερικών υδάτων να επεκταθεί η όρος του Αλιέα έτσι ώστε ένα κράτο ένα μέλος να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα ορισμού αυτού του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα. Πάμε στο 6. Ο ορισμός του αλιέα, όπως αναφέρεται εδώ, καλύπτει μόνο τη θαλάσσια αλία και δεν λαμβάνει υπόψη του ε, ορισμός ούτε την αλία εσωτερικών υδάτων, ούτε ε, την ε, υδατοκαλλιέργεια, κυρίως ε, στις περιπτώσεις όπου οι αλληλείς δεν χρησιμοποιούν αλληλεπτικά σκάφη και αυτό όμως δεν συμβαδίζει με τις ε, τρέχουσες εξελίξεις ε, που είναι η ενίσχυση κυρίως των υδατοκαλλιεργιών και των, της αλλήλειας εσωτερικών υδάτων αυτό ως εναλλακτική λύση στη θαλάσσια λία. Αυτή τη στιγμή η διατύπωση ως έχει δεν περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη του αλληλευτικού σκάφους ή τους ε, διαχειριστές ε, εσωτερικών υδάτων ή τους ε, συνειδιοκτήτες σκαφών και τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των υδατοκαλλιεργιών. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω η τροπολογία μου η 484 να στηριχτεί. Η δεύτερη τροπολογία είναι η 705. Θέλω να αφαιρθώ στην 705. Η κοινή διαχείριση θα διασφαλίσει τα ελάχιστα κονδύλια τα οποία ε, θα διατίθενται σε όλα τα κράτη-μέλη και τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προαχθεί η ολοκληρωμένη αλληλευτική πολιτική. Πρέπει λοιπόν να προάγουμε ενέργειες ε, που θα έχουν απήχηση σε όσο δυνατόν περισσότερους αλληλείς ε, και αυτά μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον υπάρχει συνδιαχείριση των κοντιλίων. Μόνο με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς ε, να επεκτείνει τον κατάλογο των αποδεκτών, των δικαιούχων, οι οποίοι θα έχουν ε, εμπειρία στην άσκηση των ε, καθηκόντων τους. Τώρα, όσον αφορά την κατάτμιση σε διάφορα στοιχεία σε σχέση με την ολοκληρωμένη αλληλευτική πολιτική, θεωρώ ότι αυτά μπορούν να οριστούν όταν όλα τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η τελευταία τροπολογία στην οποία θέλω να φερθώ, η 868 και η 869. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία εδώ είναι η ιστορική, ο ιστορικός επιμερισμός και απορρόφηση των κονδυλίων. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της κοινή ελεκτικής πολιτικής σε όλα τα κράτη-μέλη και για διάφορες περιόδους. Από την άλλη, με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατόν για μας να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα χρήσης ε, των κονδυλίων. Επίσης, κονδύλια θα πρέπει να δίδονται και στην εσωτερική αλληλεία και στο δυναμικό που περιλαμβάνει η, η, περιλαμβάνουν οι υδατοκαλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, περιορισμοί και οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν εναλλακτική λύση όταν πρόκειται για προϊόντα αλίας. Αν ε, θέλετε να μιλήσει πρώτος και ο συγητής μου και μετά εγώ. Θέλω το λόγο όμω. Πώς θα μου παλάβρα, κύριε Τόρβαλτ. Ο λόγο του κύριο Τόρβαλτ, λοιπόν. Είχα μια πιο μακροσκελή παρέμβαση ετοιμάσει, αλλά μια και ο πρόεδρος μας είπε να περιοριστούμε. Ε, θα παραλείψω ένα κομμάτι της. Νομίζω ότι καταρχήν ότι η πρόταση Κομισιόν ήταν καλή. Έχω μιλήσει με τον κύριο Καντέκ και νομίζω ότι ε, έχουμε δυνατότητα να συντάξουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση ως Επιτροπή. Το πολιετές νομικό πλαίσιο πιστεύω ότι συνδέεται αδιάρρηκτα με τον βασικό κανονισμό και με τα, τις ε, μέγιστες αποδόσεις, βιώσιμες αποδόσεις. Νομίζω ότι ε, ήδη έγινε λόγος γι' αυτό. Ε, τώρα, το καινούργια σκάφη σε σχέση με την ε, ε, διάλυση σκαφών. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Γνωρίζω ότι η μέση ηλικία των σκαφών μας είναι περίπου 27-28 έτη. Ξέρω ότι τα, ε, τα φιλανδικά σκάφη, ε, οι τράτες είναι σημαντικά πιο γερασμένα. Οι φιλανδικές τράτες παραδοσιακά ήταν η οικογενειακή διοκτησία, τώρα όμως έχουν σημαντήσει εταιρείε, οι οποίε εταιρείε εξαγοράζονται από στονικά συμφέροντα. Διατηρούν την φιλανδική σημαία όμως. Δεν γνωρίζουμε αλλά πιστεύουμε ότι ε, κάνουμε με κοινοτικά χρήματα, ε, σπαταλούμε κοινωτικά χρήματα για να κάνουμε τις εστονικές εταιρείε ικανές να αγοράσουν φιλανδικά σκάφη, γυρασμένα φιλανδικά σκάφη. Δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς λειτουργούν οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Θα πρέπει να το δούμε. Δεν θέλουμε χρήματα των φορολογουμένων να ε, προοριστούν στην αύξηση των ελευμάτων. Μαζί με τον Κρίς και τον κύριο Βάιεν έχουμε υποβάλει συγκεκριμένες τροπολογίες για αυτό το θέμα. Έχουμε επίσης ένα άλλο κοινό θέμα. Έχουμε μιλήσει για τα γυρασμένα σκάφη, αλλά έχουμε και τους γυρεούς αλείς, τους ηλικιωμένους αλείς. Είναι ένα θέμα κοινό για τις ε, βόρειες χώρες, ε, τις σκανδιναβικές χώρες και από ό,τι φαίνεται και για την Πολωνία. Έχουμε έναν πληθυσμό αλλιών πολύ ηλικιωμένο. Η πλειοψηφία τους είναι άνω των 50, κοντά στα 60. Πολύ σύντομα θα έχουμε συνταξιούχους να αλλιεύουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να έλξουμε και πιο νέους στο επάγγελμα. Δεν είναι εύκολο όμως. Όταν ταυτόχρονα προσπαθούμε να περιορίσουμε την υπεραλίευση. Ε, πολλά, άρθρα πολλά άρθρα υπάρχουν για την του καλλιέργεια. Θα πρέπει να δούμε την του καλλιέργεια. Έχουμε υποβάλει πολλές τροπολογίες για αυτό το ζήτημα. Μετά, κυρώσεις και παράνομη λατρεία και αναρχιαλία. Η αρχή της αιρεσιμότητας ε, είναι πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζεται. Δυστυχώ όμως η εφαρμογή στο παρελθόν δεν ήταν όπω θα έπρεπε, εξίσου αυστηρή. Πολύ συχνά δεν υποβάλλονται τα ε, στοιχεία, τα δεδομένα που είναι απαραίτητα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ε, παράνομης ε, λαθρέα και ανάρχης αλίας μαζί με τα κράτη-μέλη και στα υδάτα των κρατών μελών. Αυτά. Bien, gracias. Continuar. Συνεχίζουμε. Ο κ. Ντέιβις έχει το λόγο πλέον. No vamos a ver, voy a aclarar una cosa. Να διευκρινίσω το εξή. Δεν είχα δώσει ε, το λόγο εξ αρχής στους σκιώδης ηγητές, γιατί έχουμε ξεφύγει από τους, ηγητές, από τους ηγητές. Έχουμε πλέον τις ε, τροπολογίες των μελών, γι' αυτό το λόγο δεν έδωσα πρώτα το λόγο στους σκιώδης ηγητές, όπως το έκανα στην προηγούμενη μας συνεδρίαση, που η συζήτηση περιορίστηκε κυρίως στις ε, τροπολογίες και στη γνώμη των σκιωδών ηγητών. Τώρα όλα τα μέλη έχουν υποβάλει, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροπολογίες. Έχετε το λόγο. Καταρχήν μια ερώτηση προς εσάς και τη γραμματεία, Πρόεδρε. Αυτές οι τροπολογίες που σχετίζονται με τον βασικό κανονισμό, τι θα γίνουν. Αυτές οι τροπολογίες θα καταπέσουν ή θα διατηρηθούν. ε, ε ο ακούγοντα τον εισηγητή βλέπω ότι υπάρχουν, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό παρανομαστής, από, πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Ε, είμαστε υπέρ τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων, θέλουμε να υποστηριχθεί, ε, να χρηματοδοτηθεί η συλλογή δεδομένων, θέλουμε μεθόδου έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η απαγόρευση των απορρίψεων θα εφαρμόζεται σωστά μέσω επιλεκτικών εργαλείων ε, καλύτερη εμπορία και διάθεση ψαριών που παλιότερα ενδεχομένω θα σαπίζανε στην ηχθιόσκαλα. Δεν το θέλουμε αυτό. Ε, το θέμα των σχεδίων διαχείρισης, το έθιξε ο εισηγητής, ε, πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις ε, πριν το, την επεξεργασία τους ε, και ίσως θα χρειαστεί και εκεί κάποια χρηματοδότηση. Και μετά έχουμε και τα γνωμοδοτικά συμβούλια, τα ΡΑΚ, τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια, θέλουμε να μπορούν να υποβάλουν ανεξάρτητες ε, μελέτες και ενδεχομένως θα έπρεπε να χρηματοδοτηθούν ε, και αυτές. Ε, κάποιες διαφωνίες όμως, έχω και κάποιες διαφωνίες. Ο κ. Καντέκ σωστά λέει να μην αυξήσουμε την αλληλευτική δυνατότητα, αλλά η ανανέωση του αλληλευτικού στόλου μου δημιουργεί φόβο. Γιατί στο παρελθόν ε, έχει γίνει κακή χρήση ε, χρηματοδότησης ε, για τον εξυγχρονισμό αλληλευτικών στόλων. Τώρα μιλούμε για ανταλλαγή, για αλλαγή μηχανών, κινητήρων, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως αυτό θα γίνει χωρίς να αυξηθεί η αλληλευτική ικανότητα. Μετά η διαφοροποίηση. Ο εισηγητής διαφωνεί, δεν είναι πολύ ο προπολογισμό, όμως έχουμε πολλές αλληλευτικές ε, κοινότητες ε, αλλάζει η πραγματικότητα από την άλλη μεριά. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις αλληλευτικές κοινότητες που δεν έχουν άλλες δυνατότητες. Ε, πρέπει να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Εγώ δεν θα διαφορούσα με τη χρηματοδότηση, κάποια χρηματοδότηση της διαφοροποίησης, παρόλο ότι ο προπολισμός μας δεν είναι τεράστιος και πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολύ προσεκτικά. Μετά, η μικρής κλίμακος αλληλεία θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το 80% ε, των αλλιών είναι αλλιείς μικρής κλίμακος. Ε, δεν θα πρέπει τα μεγαλύτερα ποσά να πηγαίνουν στο υπόλοιπο 20%. Γιατί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και το δικό τους μέλλον. Να σας απαντήσω αυτό που νομίζω στην ερώτηση που μου κάνατε. Ίσως ο εισηγητής ξέρει καλύτερη απάντηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ασύμβατότητα μεταξύ του να υιοθετήσουμε εμείς ό,τι έχουμε να υιοθετήσουμε και ταυτόχρονα να τρέχει και ο κανόνας βάσης. Μην ξεχνάμε ότι ε, θα έχουμε πολύ μέλλον ακόμα μπροστά μας, τροπολογίες, τριμερή διάλογο, έγκριση, ε, θα λάβουμε υπόψη ε, πολλά θέματα τα οποία ε, ενδεχομένω καταρχήν ε, θα, είναι, θα έρχονται και σε σύγκρουση μεταξύ τους. Είναι απόλυτα παραδεκτό όμω. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί πρακτικά κάποιο ζήτημα εκτό και αν ο εισηγητή ή η η έχουν αντίθετη άποψη. Ο κ. Ρωμέβα. Ευχαριστώ, αλλά και εσύ έχει πολλή δουλειά και εμείς. έχουμε δύο έγγραφα να παρακολουθούμε. Αυτό που υιοθετήσαμε στο Στρασβούργο και την θέση των Υπουργών στο Σύμβουλο Υπουργών το τελευταίο Οκτωβρίου. Ε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τι ήθελαν οι κυβερνήσεις τότε και τι θέλουμε εμείς τώρα. Το ερώτημα είναι σαφές και το είπες πολύ σωστά. Η ε, συμφωνώ από τις δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια οικονομική λογική που θα αυξάνει τις αλληλευτικές ικανότητες. Το πρόβλημα όμως δεν είναι στον τίτλο αλλά στον υπότιτλο, στα μικρά γράμματα. Πώς θα γίνει αυτό. Και ο Ντέιβις το είπε πολύ σωστά. Αν δούμε το παρελθόν της ε, ευρωπαϊκής χρηματοδότηση, βλέπουμε το αντίστροφο. Σε 10 χρόνια κάναμε το ακριβώς αντίθετο. Αυξήσαμε τις ε, ε, την αλευτική ικανότητα και την υπεραλίευση. Αυτό οδήγησε σε μείωση των ε, ε, αλευτικών πόρων, αλλά ταυτόχρονα και σε σπατάλη πόρων, οικονομικών, χρηματικών πόρων. Και νομίζω ότι οι προτάσεις που μας ανακοίνωσε έρχονται σε λίγο σε αντίθεση με το στόχο μας. Εφόσον αν μιλάμε για ε, τον εξυγχρονισμό, ναι, οκ, okay, να εξυγχρονίσουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο αποδοτικοί. Αλλά ένα από τα προβλήματα που έχουμε με τους ε, σημερινούς κινητήρες ε, είναι οι ε, που έχουμε στα συστήματα ελέγχου. Συνεπώς, αν δεν επενδύσουμε πολύ περισσότερο σε συστήματα ελέγχου, δεν θα προκύψει κανένα όφελος. Θα οδηγηθούμε απλώς σε υπεραλίευση. Λοιπόν, η προτεραιότητα δεν είναι ο εξυγχρονισμός, αλλά τα συστήματα ελέγχου. Αυτό δεν νομίζω ότι το ε, αντιμετωπίζει ορθά στην έκθεσή σου. Δεύτερον, όταν ψηφίσαμε την έκθεση, ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις ε, ενισχύσεις σε ε, τομείς ε, που αλλιεύουν με τρόπο πιο βιώσιμο και πιο κοινωνικά και που είναι πιο πολύ συνδεδεμένα με την κοινωνία. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς τους τομείς αλλίας Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια τροπολογία το 291 Αυτό πρέπει να μπει στον κατάλογο. Δηλαδή να προωθήσουμε τα επιλεκτικά εργαλεία, την αλία μικρής κλίμακας, αυτή εν πάση την αλία που είναι πιο κοντά στις παράκτητες κοινότητες και να αφαιρέσουμε από το σύστημα ορισμένες ε, δραστηριότητες ε, που αποτελούν κίνδυνο γενικότερα για την αλία τα αποθέματα και προφανώς και για την συνολική ε, αλία. Τρίτο σχόλιο, και θα περιοριστώ σε αυτά, θα γίνει πιο λεπτομερή συζήτηση την Τετάρτη. Ε, πάντοτε γίνεται συζήτηση ε, για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Πώς μπορούμε να επενδύσουμε σε θέματα υγείας και ασφάλειας ε, στα σκάφη. Ναι, ναι, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις σε συνδυασμό με ε, δέσμευση των κρατών μελών να μειώσουν την αλευτική τους ικανότητα και παρακολουθώντας την αλευτική ικανότητα, τη συνολική αλευτική ικανότητα. Δεν έχουμε βέβαια καταλήξει σε ε, ένα ορισμό της αλευτικής ικανότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα καταλήξουμε. Θα πρέπει να αναλυθούν ε, Δεσμεύσει μείωση τη αλληλευτικής ικανότητα, γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν οι ε, ενισχύσεις. Μόνο αν υπάρχει μόνο αν υπάρχει μια τέτοια σαφή δέσμευση, ε, θα πρέπει να δοθούν ενισχύσεις για την ασφάλεια, την υγεία κλπ. Ευχαριστώ.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 Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Καντέκ ε, για τη δουλειά του. Ε, πραγματικά είμαι πολύ εντυπωσιασμένη με το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που κατέθεσε στους Κιώδης, που ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε έχουμε προσπαθήσει σε άλλες επιτροπές. Θα προσπαθήσω λοιπόν να κρατήσω αυτές τις ημερομηνίε. Η αντίδρασή μου σε αυτές τις περίπου 3.000 ε, τροπολογίες, όπως και άλλοι, είναι ότι δεν μπόρεσα να τις δω όλες ε, διεξοδικά, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Επέλεξα λοιπόν κάποια βασικά θέματα και από ό,τι φαίνεται έχει αλλάξει τώρα η κατάσταση από ό,τι όταν ήμασταν στο Στρασβούργο πριν από τρεις εβδομάδες, γιατί τώρα εξετάζουμε ε, το πώς θα λειτουργεί αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο σε σχέση με την κοινή ελευτική πολιτική. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί η βασική μας προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να χρησιμοποιούνται σωστά τα κονδύλια για να ε, εφαρμόζεται και η κοινή ελευτική πολιτική. Τα κονδύλια είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με ε, τα κονδύλια τα οποία χορηγούνται για την περιφερειακή ανάπτυξη και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι το Ταμείο αυτό το Ευρωπαϊκό Αλίας θα το χρησιμοποιούμε και τα κονδύλια του για την κοινή ελευτική πολιτική και όχι για άλλους ε, τομείς. Διότι ε, όταν μιλάμε για ενεργεία εκεί υπάρχουν άλλα ταμεία και έχουμε τη συμφωνία ότι αυτά τα κονδύλια θα μοχλεύονται ίσως πιο συγκεκριμένα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Ελλάς Υποθέσεις για την ανεργία, παραδείγματος χάρη. Ε, αυτό είναι προτεραιότητα για μένα. Εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιηθούν κονδύλια για την βιώσιμη ανάπτυξη, την αηφορία αν θέλετε, ε, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί από εμάς αγωνίουσαμε το να περάσει το μήνυμα στους αλληλείς ότι οι προτάσεις επί των οποίων ψηφίσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες είναι ε, υλοποιήσιμες. Να ισχύει λοιπόν αυτό όχι να δίδονται χρήματα απέναντι σε επιλεγμένα εργαλεία, αλλά και για προς την κοινωνία, για τη συγκέντρωση δεδομένων, για να διασφαλίσουμε ότι αφού θα έχουμε το σωστό εξοπλισμό, θα χρησιμοποιούμε και τα στοιχεία που θα έχουμε για να επιτύχουμε την ε, αηφορία. Βλέποντας λοιπόν τις συγκεκριμένες ε, τροπολογίες, Αναφέρομαι στις πάυσεις, ε, στις ε, προσωρινές ε, απαγορεύσεις. Κοιτάξτε, το να σταματήσει κανείς προσωρινά να λιεύει, αυτό μετά από συγκεκριμένα ερευνητικά στοιχεία πρέπει να καθιερωθεί. Αυτό σημαίνει βιώσιμη αλία. Και δεν νομίζω ότι κάθε φορά ε, να χορηγούμε επιδοτήσεις ε, όταν υπάρχει μια προσωρινή πάψη. Γιατί η επιστήμη έχει αποδείξει ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η αλία στο μέλλον και δεν πρέπει να χορηγούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα επιδοτήσεις για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Ε, θα συζητήσω με τον Ραούλ και συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι ε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό λοιπόν θα μου επιτρέψει να επανέλθω αργότερα όταν θα έχω εξετάσει λεπτομερώς όλες αυτές τις τροπολογίες. Στίβενσον, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι ο Άλαν Καντέκ ε, επέδειξε μεγάλο τάρος με τη δουλειά που έκανε έχουμε τους άθλιους, τους περίφημους, το περίφημο αυτό musical και μετά από την εξέταση όλων αυτών των τροπολογιών νομίζω ότι θα μπορούμε εμείς να ισχυριστούμε ότι είμαστε οι άθλοι. Συμφωνώ με αυτά που είπε η προλαλήσασα ότι τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τις Ελλάς Υποθέσεις είναι πολύ περισμένα και γι' αυτό πρέπει να διοχετεύονται στο σωστό χώρο και στο σωστό σκοπό. Ε, ψηφίσαμε για το ε, CCTB ε, νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων ε, διαχείρισης, κάτι που αναφέρατε στις αρχικές σας παρατηρήσεις, Αλέν, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που ε, πρέπει να το στηρίξουμε. Συμφωνώ με την Τζούλη ότι χρειαζόμαστε καλύτερα ε, επιστημονική τεκμηρίωση και σε αυτόν τον τομέα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Επίσης πρέπει να συμφωνήσουμε και για την χορήγηση κονδυλίων για την πάυση λειτουργίας μονάδων, για τον παροπλισμό τους. Ε, πραγματικά δαπανίσαμε δισεκατομμύρια κατά το παρελθόν για τον παροπλισμό μονάδων, ε, προσπαθώντας να απελευθερώσουμε ε, ικανότητες και αποτύχαμε. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν όλα αυτά τα κονδύλια και αποτύχαμε και η Κομισιόν λέει ότι δεν θα πρέπει να ξανακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Θα πρέπει να έχουμε τις ε, μεταβιβάσιμες αλληλεκτικές ε, παραχωρήσεις. Ε, αυτό το συζητήσαμε στο Στρασβούργο και γι' αυτό λοιπόν η αγορά η ίδια θα αποφασίσει μόνη της για το μέγεθος της αλληλεκτικής ικανότητας εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να στηρίζουμε μη παραγωγικές μονάδες. Αν μία μονάδα ε, παρουσιάζει ζημιά και αυτό μόνιμα, τότε όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να κλείσει η μονάδα αυτή. Συμφωνώ με τον Chris Davis ε, που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισμένα κονδύλια για τη διαφοροποίηση. Νομίζω αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε με τα διαρθρωτικά κονδύλια έτσι ώστε να βοηθήσουμε κυρίως τους τόλους μικρής κλίμακας ένα κομμάτι των ε, κονδυλίων να τα διοχετεύουν στην τουριστική ε, βιομηχανία, δηλαδή στην μετατροπή λιμένων μικρής κλίμακας που η κατασκευή τους είναι πολύ δαπανηρή, αλλά με τη βοήθεια των διαρθρωτικών κονδυλίων μπορούμε να πετύχουμε κάτι, τέτοια, τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι εφικτό. γιατί τη συντατοκαλλιέργεια συμφωνώ με τον κύριο Βαλέσα. Ε, πράγματι, ε, στα θαλάσσια προϊόντα στην Ευρώπη είμαστε αυτάρκης κατά 40%, άρα οι εισαγωγέ μας ανέρχονται στο 60%. Αυτό όμως δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να επεκτείνουμε ουσιαστικά τον αλληλευτικό μας τομέα στην Ευρώπη και αυτό προϋποθέτει επενδύσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι από όλα ένα σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια για να τα δαπανάμε για τον εξυγχρονισμό του στόλου. Μπορούν να δοθούν κάποια περιορισμένα κονδύλια για να εξυγχρονιστούν οι κινητήρες. Είπαμε ότι τα σκάφη άνω των 10 μέτρων, ε, αυτά ίσως μπορούν να χρηματοδοτηθούν με κάποιο περιορισμένο βέβαια τρόπο. Για τον ε, στόλο της ε, μικρής ε, κλίμακας, εάν διατηρηθούν οι ίδιοι οι κινητήρες και αυτούς, και αυτόν μπορούμε να τον ισχύσουμε αυτό το στόλο. Αλλά όταν μιλάμε για τον εξυγχρονισμό γενικά των ηλεκτρικών σκαφών, μην ξεχνάτε ότι δαπανίσαμε εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ με το παλιό σύστημα, μετατρέποντας τα σκάφη και ανανεώνοντας τους στόλους, αλλά τα σκάφη αυτά σε πολλά κρατημέλη εξακολουθούν να είναι νιολογημένα με την αρχική τους μορφή. Άρα δηλαδή πρέπει ε, να εξετάσουμε την νιολόγηση και να πάμε πίσω 20-30 χρόνια. Δόθηκαν πολλά κονδύλια για τον πλήρη εξυγχρονισμό των στόλων. Εγώ δεν θα ξαναπέσω σε αυτή την παγίδα δεν θα πρέπει ο πλήρης εξυγχρονισμός να διεισδύσει στην συζήτησή μας. Υπάρχουν λοιπόν αυστηρές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κύριε Πρόεδρε και κατά την άποψή μου πάνω σε αυτές τις παραμέτρους πρέπει να επικεντρωθεί η συζήτηση. Η κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισήγητη. Πρώτα απ' όλα θα ασχοληθώ με το θέμα της ε, αλίας μικρής κλίμακας. Πιστεύω ότι θα πρέπει για αυτή την αλία να υπάρξει συνενετική λύση. Έχω εγώ μία σχετική τροπολογία, αλλά συμβαστική λύση θα πρέπει να είναι όποια είναι, αλλά πρόκειται για συμβαστική λύση. Δεν είμαι όμως υπέρ αυτών που λένε ότι κάθε χώρα κάνει ό,τι θέλει. Πιστεύω ότι ο ορισμό θα πρέπει να είναι ενιαίος, θα πρέπει να βελτιωθεί ο παρόν ορισμός, διότι πιστεύω ότι αν κάνει κάθε χώρα ό,τι θέλει, τελικά μπορούμε να οδηγηθούμε σε διακρίσει μεταξύ αλλιευτικών στόλων ε, κρατών μελών που αναπτύσσουν τι αλληλευτικές δραστηριότητε στις ίδιες περιοχές. Άρα αντί να κάνουμε θετικές διακρίσεις, θα κάνουμε το αντιθετικό. Είμαι λοιπόν εγώ υπέρ ορισμού. Ενό ορισμού, όποιο και να είναι αυτό όσον αφορά λοιπόν την αλληλεία μικρή κλίμακα. Όσον αφορά του στόχου και τι προτεραιότητε, πιστεύω ότι στην πρόταση τη Επιτροπή, εκτό από την υδατοκαλλιέργεια, έχει ξεχαστεί και η μεταποιητική βιομηχανία. Και θα πρέπει να τη συμπεριλάβουμε εδώ, διότι είναι η μεγάλη ξεχασμένη στην μεταρρύθμιση. Τώρα, στο άρθρο 13 και στις μη επιδοτούμενες δραστηριότητες. Είμαι κατά των νέων κατασκευών. Για ποιο λόγο. Πρώτα απ' όλα, διότι νομίζω ότι οπισθοδρομούμε αυτόν τον τρόπο. Δεύτερον, διότι παρά το γεγονός ότι λέμε ότι θα υπάρξουν νέα σκάφη, και αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ικανότητα, αυτό είναι λαθασμένο, Διότι στο παρελθόν είδαμε ότι αυξήθηκε η ελευτική ικανότητα με αυτόν τον τρόπο. Άρα δεν είμαι υπέρ των νέων ε, ε, κατασκευών και νέων πλοίων σε καμία περίπτωση. Τώρα, θα ήθελα να πω το εξή. Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ υπήρχε ένα πρότυπο διαχείρισης, το οποίο περίφθη, αλλά σε αυτό το πρότυπο διαχείρισης είχαμε ως θετική επίπτωση την μείωση της αλληλευτικής ικανότητας. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε λοιπόν, δεν εγκρίθηκε αυτό, όπως είδαμε για τα θέματα των μεταβιβάσεων αδειών είδαμε ότι χρειάζεται πραγματικά τώρα να δοθεί κάποια ενίσχυση για την απόσυρση κάποιων, για την βάση λειτουργία. Και ο αλλιευτικό στόλο πιστεύω ότι δεν έχει δυνατότητα από μόνη τη να μειωθεί, άρα χρειάζεται κάποιε ενισχύσει, κάποιε επιδοτήσει. Κατά συνέπεια, είμαι υπέρ αυτή τη ενίσχυση όσον αφορά την προσωπική, την προσωρινή ε, πάυση κάποιων δραστηριοτήτων. Ξέρω ότι κάποιοι το επέκριναν, αλλά ποιος μπορεί να επικρίνει το ότι κάποια στιγμή προσωρινά γίνεται μία πάυση δραστηριοτήτων όταν ε, υπάρχει ρήπανση στην θάλασσα. Ξέρουμε, το έχουμε ζήσει πολύ και ξέρουμε ότι κάποιες επίγουσες καταστάσεις δικαιολογούν αυτή την ενίσχυση σε περίπτωση ε, απότομης πάυσης λειτουργίας. Τώρα, όσον αφορά την αποθεματοποίηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπήρχε ήδη στον ε, έκθεση την οποία έκανε ο κύριος Στίβερσης για τον ε, κανονισμό. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν την ενίσχυση για την αναποθεματοποίηση να την απορρίψουν. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να, συνεχιστεί. Δεδομένου ότι είναι το μοναδικό ε, θέμα το οποίο είναι μία από τις διασφαλίσεις που προσφέρουμε. Όλες οι άλλες οι ενισχύσεις καταργήθηκαν. Ένα άλλο θέμα. Και αυτό αντικατοπτρίζεται σε κάποιες τροπολογίες. Το θέμα χρηματοδότησης και του του 1, 2, 3%. Εάν σεβόμαστε το χρονοδιάγραμμα, ναι ή όχι, στα πλαίσια του προγραμματισμού. Εγώ, ακόμη και αν είμαι μόνη μου, θα ήθελα να συνεχίσει η ενίσχυση της αποθεματοποίησης, να μην ε, μειωθεί και να δούμε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα πώς θα την ε, ε, δώσουμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της διαφοροποίησης. Η Κομισιό τα θέλει όλα εκτός του αλληλευτικού τομέα. Άλλοι μόνον. Εγώ είμαι υπέρ και για τον αλληλευτικό τομέα και εκτός. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιοριστούμε σε ένα ή στον ένα ή στον άλλο τομέα της παραγωγής. Νομίζω ότι αιτιολογείται απολύτως αυτή η αρχή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε τη διαφοροποίηση. Αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις που θέλω να κάνω. Σταματώ. Ευχαριστώ κύριε Ρόντουστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον συνάδελφο κύριο Καντέκα. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει το να καλείται κανείς να χειριστεί τόσες πολλές ε, τροπολογίες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η συνεργασία με τους ε, σκιώδεις ηγητές είναι τόσο αγαστή. Ε, σου είμαι ευγνώμων αγαπητέ αλλά το, για το γεγονός ότι παίρνει το βασικό κανονισμό ως τη βάση εκείνου πάνω στο οποίο θα διαμορφωθεί το Ευρωπαϊκό αυτό Ταμείο. Και πολύ καλά κάναμε και καθυστερήσαμε την έκθεση αυτή για να μπορέσουμε να πάρουμε ως βάση το βασικό κανονισμό. Ε, πράγματι ε, δίδει μεγάλη σημασία στην επιλεξιμότητα και ο έλεγχος μοιάζει να είναι πολύ σημαντικός για, σένα. Με τους συναδέλφους που πήγαμε στην Ιρλανδία ε, διαπιστώσαμε ότι πραγματικά όσο έλεγχο και να ασκούμε, ορισμένοι σε αποδεικνύονται τόσο εφάνταστοι που καταφέρνουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Τέτοια φαντασία δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια ε, εδώ στη δική μα θέση. Αυτό που κάνουν αυτοί στον Ατλαντικό ούτε να το σκεφτούμε δεν μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν ο έλεγχο πρέπει να είναι πολύ σοβαρό και να διατυπώσουμε τα μέτρα μα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να υπάρχουν ω το δυνατόν λιγότερα παραθυράκια. Ε, Βεβαίω αυτό δεν ισχύει για την πλειοψηφία των αλλιέων που γνωρίζω ότι εργάζονται ε, νομότυπα. Δεν συμφωνώ με αυτό που λες Αλέα ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ανταγωνιστικότητα δηλαδή να ε, επιδοτούμε τους αλλοίς όταν πάβουν την δράση τους, όταν πάβουν να ασχολούνται με την αλία. Κοίταξε και στη Γεωργία πάρα πολλοί Γεωργοί εγκατέλειψαν τη Γεωργία και πρέπει να τους δίδεται η δυνατότητα της ε, κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης. Ε, να το τονίσουμε αυτό, ότι αν οι αλληλείς επιθυμούν και να υπογραμμίσουμε ότι επιθυμούν να αλλάξουν επάγγελμα, εμείς θα τους ε, χρηματοδοτούμε. Άρα πρέπει να προβλέπουν κονδύλια. Όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των στόλων, είναι ένα δύσκολο θέμα το έχουν θίξει πάρα πολύ. Κατά την άποψή μου η γύρανση δεν είναι καθοριστικό κριτήριο. Για μένα είναι σαφές ότι οπουδήποτε υπάρχει πλεονάζουσα αληθική ικανότητα μπορούμε να προβλέπουμε την ε, διάλυση των σκαφών. Και όπου δεν υπάρχει πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα, εκεί μπορούν να υπάρξουν νέα σκάφη, αλλά μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Πώς ορίζεται η πλεονάζουσα αλληλευτική ικανότητα, μέχρι τώρα δεν το έχουμε ορίσει με σαφήνεια. Και δυστυχώς η Κάρμεν έχει επίσης δίκιο, δεν έχουμε ορίσει τι είναι η μικρή και παραδοσιακή αλία. Εγώ είχα ελπίσει με την έκθεση Φερέιρα να επιτύχουμε λογικούς ε, ορισμούς, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Έτσι λοιπόν, ε, σε αυτά τα δύο θέματα υπολείπονται ακόμα πάρα πολλά, αλλά σε επίπεδο αρχής εγώ τάσομαι υπέρ της διάλυσης σκαφών όπου προκύπτει πλεονάζουσα αληθική ικανότητα. Και ανανέωση στόλων μόνο εφόσον δεν υπάρχει πλεονάζουσα ικανότητα, βεβαίως τη σωστή διατύπωση πρέπει να την αναζητήσουμε. Η ε, κυρία Πατρά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να πω ότι όταν διάβασα την πρόταση επιτροπή για πρώτη φορά σε σχέση με το ΕΤΑ, σχημάτισα την εντύπωση ότι πρόκειται κυρίως για ένα έγγραφο που αφορά την έξοδο από το επάγγελμα και αυτό με απασχόλησε πάρα πολύ. Όταν ε, σκέφτομαι ότι εδώ κυρίως θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, λέξεις να αλλιεύουμε καλύτερα. Το είπε αυτό ο εισηγητής και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και να τον συγχαρώ για την ε, εργασία του. Θα ήθελα να πω και εγώ ότι και εγώ βρίσκομαι σε σχεδόν πλήρη συμφωνία με όλα αυτά τα οποία ανέφερε και εξήγησε ο εισηγητής. Όντως πιστεύω ότι η λέξη κλειδί για μας θα πρέπει να είναι καλύτερη αλληλεία και να δώσουμε τη δυνατότητα στους αλείς, όχι να χρειάζεται να ψαρεύουν περισσότερο για να έχουν καλές αποδοχές, αλλά να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν με καλύτερη κατάρτιση. Με κατάρτιση των αλλιέων, ακόμη και για να μπορούν να επεξεργάζονται καλύτερα τα αλλιεύματά τους, ώστε να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα να τους μάθουμε ότι δεν χρειάζεται να αλλιεύουν περισσότερο και να μην θέτουν σε κίνδυνο τους αλλιευτικούς πόρους και να μάθουν ότι αυτό δεν έχει κανένα όφελος, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις και να δώσουμε τα μέσα και τις συνθήκες για να μπορούν να αλλιεύουν όλο και καλύτερα οι αλλιείς. Πρώτα απ' όλα, στοιχηματίζοντας τη σωστή κατάρτιση και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφές, Δεύτερον, ώστε να γίνει το επάγγελμα τη αλλιέως ένα αξιόπιστο επάγγελμα. Δύσκολα θα μπορέσουμε να προωθήσουμε την ανανέωση του επαγγέλματος εάν δεν μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους νέους, περισσότερους νέους ανοιχτούς στην σημερινή πραγματικότητα της μεταποίησης των αλλιευμάτων, με δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος που δεν έγιναν τις προηγούμενες γενιές. Νομίζω ότι αυτά είναι πρωτερχικά σημασία θέματα για να αντιμετωπιστεί η σημερινή πραγματικότητα και να αλλιεύει καλύτερα ο αλλιέας σήμερα. Πιστεύω όμως ότι γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους αλλιείς να κάνουν μια δραστηριότητα πιο αποδοτική. Διότι αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι η ποσότητα, αλλά η απόδοση. Διότι ο Αλιέας δεν θα υπεραλλιεύει εάν έχει την δυνατότητα να έχει καλή απόδοση των ε, πολίσεων, των ε, αλιευμάτων που με τον καθημερινό του μόχθο αλλιεύει. Θα πρέπει επίσης να μπορέσουμε να προωθήσουμε την επιστημονική ε, έρευνα, πραγματογνωμοσύνη, την ενοποίηση των μεθόδων που ακολουθούνται, διότι όλα τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους και για να έχουμε μία ισότιμη κατάσταση για όλους, τα πρότυπα θα πρέπει να είναι ενιαία και συγκρίσιμα για όλους. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε σε θέση τα δεδομένα που συλλέγονται στις διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούμε να τα συγκρίνουμε για να έχουμε μία προσέγγιση οικοσυστημική. Πράγμα το οποίο απαιτεί η ανάγνωση να γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Επίσης, θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην ε, ε, εμπειρική αλληλεία για να μειωθούν και η πίεση που ασκείται στα αλλιεύματα εφόσον μιλούμε για τις προσωρινές μεταβιβάσεις άδεια αλληλείας και τις παραχωρήσεις, όπως και η Κάρμεν και εγώ το υποστηρίζω αυτό και είμαι εντελώς αντίθετη σε επιχειρήματα ότι αν δεν μπορεί κανείς να αλλιεύσει δεν αλλιεύει, διότι μιλούμε για επαγγελματίες που αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχουν καμία δυνατότητα αλλιεύσης. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα σημαίνει για αυτούς ότι ε, δεν θα φάω και αυτό το μήνα, θα φάω τον επόμενο αν μπορέσω να αλλιεύσω. Νομίζω ότι αυτό είναι εξωπραγματικό και θα πρέπει να το αφήσουμε σε επιχείρημα κατά μέρο. Επίσης μου φαίνεται ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε με αξιοπρεπή την έξοδο κάποιων αλλίων από το επάγγελμα και αυτή η έξοδος θα πρέπει να γίνει με τρόπο που θα αμβλύνει την πίεση στα αλλιεύματα. Κάτι άλλο το οποίο το ήθελα οπωσδήποτε να αναφέρω είναι η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός του αλλιευτικού στόλου. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να συνοδεύεται και με τις βελτιώσεις που θα γίνουν στους λιμένες αλλιεύσεις, ώστε να περιέχουν ε, καλύτερη ε, διοικητική υποστήριξη και μεγαλύτερη ασφάλεια. Διότι πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι αλληλευτικοί στόλοι που εξυγχρονίστηκαν, άλλοι όχι. ο Πορτογαλικός αλληλευτικός στόλος δεν ε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι θα πρέπει ε, όλα τα πράγματα να τα δούμε με τρόπο ορθολογιστικό και μετρημένο. Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε εξάλλου για τον εξυγχρονισμό του αλλιευτικού στόλου ε, μία ε, άποψη, ας κάνει ο καθένας ό,τι επιθυμεί, αλλά να έχουμε μία ορθολογιστική άποψη. Και η ασφάλεια, επαναλαμβάνω, εδώ είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Η βελτίωση των λιμένων ούτως ή άλλως και της δυτικής υποστήριξης στους λιμένες είναι πολύ σημαντική επίσης από τη στιγμή που μιλούμε για περιορισμό των απορρίψεων. Εγώ είμαι από μια εξόχως απομακρυσμένη περιοχή η αλία στα εννέα νησιά των Αζωρών είναι κάτι που μπορώ να σας εγγυηθώ ότι δεν επιτρέπει ε, σε κανένα από αυτά τα νησιά να διαχειριστούμε το θέμα των απορρίψεων. Δεν υπάρχει σε κανένα από αυτά τα εννέα νησιά να ξέρουμε τι γίνεται με τις απορρίψεις. Και βεβαίως Μιλώ για μηδέν μεταποιητική βιομηχανία που θα χειριστεί αυτές τις απορρίψεις. Θέλησα να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Ε, γι' αυτό ανέφερα μόνο τα σημαντικά θέματα. Υποστηρίζω αυτά τα οποία ελέγχθησαν. Συμφωνώ με τους συναδέλφους. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι αυτή η υποστήριξη της μικρής κλίμακας αλίας είναι ακόμη πιο σημαντική για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές και όταν μιλούμε για ένα νησί με 300 κατοίκους που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αλληλεία, δεν θα αφαιρέσω τη δραστηριότητα από τους κατοίκους της, διότι μιλούμε για περίμωση. Τώρα, για το θέμα της αποθεματοποίησης. Συμφωνώ με αυτά που είπε η Κάρμεν και εγώ συμφωνώ ότι το τελευταίο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αυτό για να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε και σε σχέση με τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν θα ήθελα να προσθέσω και το εξή. Η αποθεματοποίηση επιτρέπει την επανεισαγωγή των αλλιευμάτων ε, στην αγορά όταν υπάρχει μικρότερη προσφορά ή μεγαλύτερη ζήτηση. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε αυτό το θέμα, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με καλύτερη παραγωγικότητα. Τώρα, όσον αφορά την ενίσχυση για την εκμετάλλευση και την εμπορία, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν υπήρχε στην πρόταση της Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επανεισαχθεί. Υποστήριξη στην υδατοκαλλιέργεια είναι ζωτική σημασία για την αλία και για την ευρωπαϊκή οικονομία και εκτός από όλα τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν θα αμβλύνει και την πίεση στην αλία. Διότι με την ανάπτυξη της υδατοκαλλιεργίας θα αμβλύνουμε περισσότερο την πίεση στην παραδοσιακή αλία. Τώρα, Όσον αφορά την λειτουργία των CCR, πιστεύω ότι είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης, της περιφερειοποίησης και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους τοπικής φορείς, τοπικούς φορείς μεγαλύτερες αρμοδιότητες. Και θα πρέπει να διαθέσουμε και μέσα για νέες αρμοδιότητες που θα τους αναθέσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ η κυρία Γκαρθία Γέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Καντέκ για την κατανόηση του. Πολλές οι τροπολογίες, αλλά σίγουρα, κύριε Καντέκ, είχατε την ευκαιρία να τις δείτε όλες μαζί ε, και να δείτε αν πράγματι πρόκειται για διαφορετικά πράγματα. Πολλές φορές ε, υποβάλλονται πολλές μεγάλους αριθμούς τροπολογιών, αλλά μιλάνε για το ίδιο πράγμα. Ε, μας είχε ζητηθεί άλλωστε να μην υποβάλουμε πολλές τροπολογίες και προσπαθήσαμε εμείς ως Ισπανική Αντιπροσωπεία να διευκολύνουμε τη δουλειά σας, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Το πλαίσιο είναι αυτό το οποίο έχει εγκριθεί στο Στρασβούργο και αυτό είναι το πλαίσιό μας και θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτό το πλαίσιο. Οι στόχοι του ταμείου σίγουρα δεν θα πρέπει να οδηγούν στην αύξηση της αλίευσης. Τούτου λεχθέντος, η χρήση του ταμείου και γενικότερα των ταμείων μπορεί να είναι όσο πλατιά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα εργαλεία, για τις αληθικές ικανότητε, για την ανάγκη της αλίας, της υδατοκαλλιέργειας κλπ. είμαστε ένα μοσαϊκό χωρών, αναγκών και πραγματικότητων. Ε, γι' αυτό λόγο πρέπει να είναι ε, πλατή, ε, ευρύ το πεδίο εφαρμογή. Είχα υποβάλει μια τροπολογία η οποία απορρίφθηκε και από την ομάδα μου για τον ορισμό της αλίας, της παράκτης αλίας και της αλίας μικρής κλίμακας. Δεν είναι δυνατόν να τον αποφύγουμε. Αλλά μου υπόψη της εκθέσεις ε, του Ελληνικού Συνεδρίου θα δούμε ότι δεν έχει γίνει σωστή χρήση αυτών των όρων ε, στην χρηματοδότηση δραστηριοτήτων. Αυτοί που έχουν πάρει τα μεγαλύτερα χρηματοδότηση είναι οι πιο ισχυροί, ε, οι πιο ικανοί να υποβάλουν πλήρη και ολοκληρωμένα σχέδια εξυγχρονισμού, διάλυσης ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα μιλούμε για διάλυση, αλλά στην πραγματικότητα αυτά τα σκάφη αντικαθίστανται από άλλα ε, πιο ισχυρά, μεγαλύτερη λευκή ικανότητα. Λάθο αυτό. Ο εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμό τι σημαίνει. Εξυγχρονισμό όχι για την αύξηση τη αλληλευτική ικανότητα. Το λέω πάντοτε αυτό. Ε, ο εξυγχρονισμό ε, έχει ως στόχο την προσαρμογή αυτών των σκαφών σε και στους καινούριους ε, χρόνους, καινούριους καιρούς, αλλά και σε πιο υγιείς συνθήκες ε, εργασίας, εν προσαρμογή ε, σε, στις, περιβαλλοντικές απαιτήσει, για παράδειγμα κινητήρες που μολύνουν λιγότερο κλπ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηρίξουμε μέσω του ταμείου αυτού όλο το τομέα της αλίας χωρίς να αυξήσουμε την υπεραλίευση. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω κάτι το οποίο έχουμε ξεχάσει, είναι ένα τομέα τον οποίο έχουμε ξεχάσει. Ε, είναι ο, ο τομέας της ε, αλίας μικρής κλίμακας. Οι μικρή αλίες, τα μικρά αλλιευτικά σκάφη ε, βλάπτονται ε, και, και όλα γίνονται εις βάρος τους και υπέρ των λιγότερων αλλά πιο ισχυρών. Δεν είναι δυνατόν να τους ξεχνάμε. Ελπίζω να το λάβετε υπόψη να δεχτείτε κάποιες από τις τροπολογίες μας. Στο άρθρο 48, συμφωνούμε με την ε, τροπολογία για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων, των γυναικών, ε, για να αποφευθούν οι διακρίσεις και επίσης ε, να καταρτιστούν και να εργαστούν και άτομα με αναπηρίες, ανάλογα βέβαια και στο μέτρο των ικανοτήτων τους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν κονδύλια που θα βοηθούν ε, τις ε, περιοχές ε, που λόγω ψηλών δικτών ανεργίας θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Υπάρχουν περιοχές που ζουν αποκλειστικά από την αλία μπορούμε να τις βοηθήσουμε με κατάρτιση έτσι ώστε να αποκτήσουν και άλλου τύπου πόρους, οικονομικούς πόρους ε, και να ασχοληθούν και με άλλες δραστηριότητες. Το κάναμε ε, με τα αυτοκίνητα, στην βιομηχανία, Τα προγράμματα που έχουμε χρηματοδότησης, αγοράς νέων, ε, λιγότερο ε, ε, αυτοκινήτων τα οποία μολύνουν λιγότερο αλλά και όχι μόνο τέτοιων αυτοκινήτων και ε, όχι μόνο τέτοιο αυτοκινήτων πολλές φορές ε, χρηματοδοτούμε και ε, πιο ρηπογόνα μεγαλύτερα αυτοκίνητα ε, και αυτό επιδότηση είναι μετά θα πρέπει να δούμε το, τη χρήση των επιστημονικών δεδομένων θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τις επιστημονικές έρευνες μία από τις τροπολογίες μας ε, λέει επίσης ότι όταν υπάρξει ε, μία φυσική καταστροφή δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τους αλληλείς στην τύχη τους. Ποιο θα μπορούσε να πει ότι θα έπρεπε του ε, αλληλεί να του αφήσουμε στην τύχη του, Γιατί αυτού και όχι άλλου οικονομικού τομεί. Μιλάμε για στόχου, δεν μιλάμε για ποσότητε, έτσι. Μιλάμε για στόχου. Μιλάμε για κριτήρια. Μιλάμε για κριτήρια επιλεξιμότητας. Είναι και αυτό ένα κριτήριο. Μετά, το τέλο η ανταγωνιστικότητα. Και η ανταγωνιστικότητα είναι κριτήριο. Γιατί το γεγονό ότι υπάρχει υπεραλίευση, υπερεκμετάλλευση. Η χρήση ε, η υπερβολική χρήση των ε, αλλιευτικών εργαλείων ε, ε, ότι δεν σημαίνει λέω ότι δεν μπορούμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα χωρίς να αυξήσουμε την υπεραλίευση. Χρειάζεται, υπάρχει περιβαλλοντική και κοινωνική αποδοτικότητα για παράδειγμα και αποτελεσματικότητα. Έχουμε τροπολογίες για όλα αυτά τα θέματα, ίσως τις βρείτε πολλές, αλλά ε, μην ξεχνάτε ότι... Ε, δεν μας δίνονται και πολλές ευκαιρίες να συμμετάσχουμε και να επηρεάσουμε τις αποφάσεις εμείς οι ευρωβουλευτές. Γι' αυτό το λόγο αξίζει να κάνετε τον κόπο να τις διαβάσετε. Οι υποφαινόμενοι ε, πολύ ευχαρίστω θα αποσύρει ω μέσα τροπολογίε αν δεχτείτε τι βασικέ. Ευχαριστώ πολύ, Ο κ. Φερέιρα. Ε, Καταρχήν ένα γενικό σχόλιο και μετά θα αναφερθώ σε κάποιες πιο συγκεκριμένες τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Η πρόταση της ε, Κομισιόν ε, μόνο με πολύ, ε, ε, πολύ λίγο αυστηρά κριτήρια μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αφορά ένα ταμείο για την αλία για τη θάλασσα. Πιο πολύ τομέα, σε διάλυση τομέα οδηγεί. Βέβαια, ο εισηγητής προσπαθεί να διορθώσει πολλές από τις αδυναμίες. Όχι όλες όμως, της αρχικής πρότασης είναι δυνατόν και απαραίτητο να πάμε ακόμα πιο μακριά στην διόρθωση αυτών των αδυναμιών, των ανεπαρκειών της πρότασης Κομισιόν. Από τις πολλές ε, προτάσεις τροπολογίας ε, που υπέβαλε η ομάδα μας, 150 περίπου, θα αναφερθώ σε ορισμένες μόνο. Σε άλλες αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την είσοδο νέων αλλιών. Έχουμε ένα τομέα που έχει γεράσει πολύ σε πολλές χώρες. Και αυτό, ε, επιστρέφοντας λίγο πιο πίσω, είναι το βασικό πρόβλημα της αρχικής πρότασης. Ότι αγνοεί πως υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία της αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολύ, πολύ διαφορετική πραγματικότητα των στόλων, των χαριστικών των στόλων, των ε, αλευτικών πόρων, των εργαλείων που χρησιμοποιούνται, των διαφόρων ειδών που αλλιεύονται κλπ. Ο κανονισμός το αγνοεί αυτό. Η, και η μέση ηλικία του στόλου είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Υπάρχει ένα όρο, αλλά υπάρχουν πολλές αποκλήσεις. Και ο κανονισμός, δυστυχώς, όπως και ο βασικός κανονισμός, αγνοεί ε, αυτή την μεγάλη ποικιλομορφία. Μίλωσα για την είσοδο λοιπόν νέων αλλιών στο επάγγελμά Το επάγγελμα, το αυτό είναι ένα πολύ σκληρό επάγγελμα και ε, απογράφουμε το θάνατο του επάγγελματος αν δεν φροντίσουμε να μπουν και, νέοι στο επάγγελμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι το έχει αντιληφθεί. Η Επίτροπος ε, πρόσφατα στην Ολομέλεια ε, είπε ότι είναι πρόθυμη να διορθώσει αυτή την αδυναμία της αρχικής πρότασης προβλέποντας ε, την υποστήριξη εισόδου νέων αλλιών. Μακάρι. Σε ό,τι αφορά τις ε, επίγες υποδομές. Και εδώ η κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και ορισμένες χώρες και ιδίω σε περιοχές αλλιές μικρής κλίμακας ε, υπάρχει μια σοβαρή και σαφής έλλειψη επίγειων υποδομών. Ε, ε, ε, λιμάνια, προβλήτες εκφόρτωσης, γενικώ υποδομές εκφόρτωσης κλπ. Δηλαδή υποδομές που θα δίνουν προσθέμενη αξία στη δουλειά του Αλία πρώτη μεταποίηση, για παράδειγμα, κλπ. Ο κανονισμός αγνοεί τελείως όλε αυτές τις ανάγκες. Ο εισηγητή διορθώνει και πολύ σωστά εν μέρη ορισμένα από αυτά τα προβλήματα. Εμείς έχουμε κάνει ακόμα περισσότερες προτάσεις. Πηγαίνω ακόμα πιο μακριά προκειμένου να γνωρίσουμε την ανάγκη να υποστηριχθούν τέτοιου είδου ε, επίγειες ε, υποδομές. λέω, σε περιοχέ ε, ε αλίας, ε, μικρής κλίμακας και για λόγους ασφαλείας, μεταξύ άλλων. Χρειαζόμαστε καινούρια αλευτικά λιμάνια. Μιλώντας για την ασφάλεια, υπάρχει και το ζήτημα της αντικατάστασης των κινητήρων. Λόγοι ασφαλείας επιτάσσουν ιδιαίτερο στην αλληλεμικές κλίμακα την αντικατάσταση των κινητήρων. Η αντικατάσταση γίνεται για λόγους ασφαλείας. Ίσως κάποιοι αγνοούν την πραγματικότητα, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν αλλοί στα ύδατά μας, άνθρωποι οι οποίοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να πάνε να ψαρέψουν, γιατί αλλιώς θα πεθάνουν τη πείνας. Έχουμε παράκτιες ε, περιοχές ε, που διέρχονται σοβαρή οικονομική και κοινωνική κρίση όπου δεσπόζει ο τομέας της ε, μικρής κλίμακας. Συνεπώς ε, υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι ασφάλειας στην αντικατάσταση των κινητήρων. Συνεπώς να εγκρίνουμε γενικές αρχές οι οποίες αγνοούν την τοπική πραγματικότητα είναι λανθασμένο κατά την άποψή μας. Θα πρέπει να διορθωθεί στην πρότασή μας. Και ό,τι αφορά τις ε, βιολογικές παύσεις, τις ε, προσωρινές πάυσεις δραστηριοτήτων. Υπάρχουν βιολογικοί λόγοι, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν γίνεται η υπεραλίευση. Μερικές φορές είναι απαραίτητο ε, σε κρίσιμες φάσεις ε, της, του, του κύκλου ζωής των αλευτικών αποθευμάτων. Αυτό αναγνωρίζεται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Τέτοιου είδους προσωρινές πάυσεις δραστηριοτήτων είναι για να εξασφαλιστούν εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αλλιών. Όμως, κατά τη διάρκεια αυτών των περίοδων, οι αλλοί θα πρέπει κάπως να επιβιώσουν. Η ασυνέχεια της οικονομική δραστηριότητα που είναι αδιάρρηκτα δεμένη με την, με την ίδια δραστηριότητα θα πρέπει ε, να ε, ε, αποζημιωθεί στους αλλοίς. Σε ό,τι αφορά τα επιστημονικά δεδομένα. Το είπε και ο εισηγητή και άλλοι. Είναι απολύτω απαραίτητο να βελτιωθεί η γνώση τη κατάσταση των αλλιευμάτων, των αλλιευτικών πόρων ή αλλιευτικέ πολιτικέ, τι οποίε καθορίζουμε αυτή τη στιγμή για τα επόμενα χρόνια, χαρακτηρίζονται από έλλειψη επαρκού γνώση τη κατάσταση των διαφόρων λευτικών ειδών ή των διαφόρων αλλιευτικών ειδών ε, ή των διαφόρων αλλιευτικών ζωνών. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα και είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει και το κόστος δεν είναι δυνατόν ε, να διαθέτουμε κοινή αλληλευτική πολιτική, αλλά μετά τα κόστη να τα σπρώχνουμε προς την πλευρά των κρατών μελών. Δηλαδή, εφόσον η αλληλευτική πολιτική είναι ε, αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει και το κόστος της συλλογή αυτών των δεδομένων. Αν όχι όλο το κόστος, θα πρέπει να αναλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος του. Τώρα η πρόταση του ε, εισηγητή είναι αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης. Δεν είναι αρκετή. Εγώ έκανα μια πρόταση ακόμα, μεγαλύτερη ακόμα μεγαλύτερης αύξησης του ποσοστού χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα λεπτό ακόμα, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, για να μιλήσω για ε, την ε, αλία ε, μικρής κλίμακας. Έχω υποβάλει έκθεση για αυτό το θέμα με συγκεκριμένε συστάσει, ορισμένε από τι συστάσει, τι υποβάλλουμε και ω τροπολογίε σε αυτή την έκθεση. Θέλω όμω να σα υπογραμμίσω την σημασία όλων των τροπολογιών των σχετικών με την αλία μικρή κλίμακας, αλλά ιδιαίτερω στην πρόταση αύξηση των ενισχύσεων λίγο παραπάνω από το επίπεδο προτείνει κομισιόν. Εμεί κάναμε μια πρόταση ορισμού που κατά την άποψή μας ε, βελτιώνει τον ορισμό της αλίας μικρής κλίμακας στο κείμενο, ε, που δεν συνάδει με αυτά τα οποία συζητούσαμε ε, στο πλαίσιο του κειμένου της έκθεσης για την αλία μικρής κλίμακας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιεί και τον όρο της διάρκειας της παλήρια. Μπορεί να βελτιωθεί λοιπόν ο ορισμό, είναι σημαντικό και πρέπει να βελτιωθεί. Έχουμε κάνει πρόταση γι' αυτό. Τώρα, για την υδατοκαλλιέργεια. Και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, ε, μεγάλη ποικιλία καταστάσεων που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θετικό ε, να υποστηρίξουμε καινοτόμε μορφές υδατοκαλλιέργεια, για παράδειγμα στην ανοιχτή θάλασσα. Αλλά αυτού του τύπου η υδατοκαλλιέργεια είναι αδύνατη σε ορισμένα κράτη-μέλη. Με δεδομένο το επίπεδο που βρίσκεται η τεχνολογία αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί σε πολλέ χώρε ε, η υδατοκαλλιέργεια ανοιχτή θάλασσα. Συνεπώ, ναι, να υποστηρίξουμε και τέτοιου είδους υδατοκαλλιέργειες, αλλά όχι μόνο αυτές, διότι μα, αν, με αυτόν τον τρόπο οι χώρες που ε, βλέπουν προς τον Ατλαντικό ωκεανό ε, δεν θα μπορούσαν να υποστηριχθούν καθόλου στην υδατοκαλλιέργειά τους. Τώρα, για τις έκτακτες περιστάσεις και τις ενισχύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σημαντικό να διαθέτουμε μηχανισμούς που θα εγγυώνται την υποστήριξη σε τέτοιους έκτακτες περιπτώσεις, φυσικές καταστροφές, το είχαμε ήδη προτείνει και στην έκθεση για την αλία μικρής κλίμακας. Ε, ο, έχουμε στον προπολογισμό μας ε, δυνατότητα, κονδύλια για να δράσουμε σε τέτοιους περιπτώσεις για τη γεωργία, γιατί όχι και για την αλία όπως και η γεωργή και η γεωργία γενικότερα είναι ευαίσθητη έναντι ε, μετρολογικών φαινομένων, καιρικών φαινομένων, φυσικών καταστροφών, θεομηνιών κλπ. Έτσι θα πρέπει να έχουμε και κάποιους παρόμοιους μηχανισμούς για την αλία. Ευχαριστώ κύριε Thank you, Chair. And... Πρόεδρε και ευχαριστώ τον, ευχαριστούμε τον Αλέν για την έκθεσή του και βεβαίως έχετε πάρα πολλή δουλειά μπροστά σας με όλες αυτές τις ε, τροπολογίες. Ο συνάδελφός μου Ραούλ ήδη ανέφερε τα σημαντικότερα θέματα για μας, για τους πράσινους, γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά πρώτα απ' όλα νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε τους αυτούς μας ε, για την ε, ψηφορία την Πέμπτη στην Ολομέλεια, όπου αποφασίσαμε ότι θέλουμε να αναμορφώσουμε τα αποθέματα σε τέτοια επίπεδα έτσι ώστε να μπορούν να ε, προσφέρουν το ανώτατο ε, βιώσιμη, την ανώτατη βιώσιμη απόδοση. Αν δείτε τη Νέα Ζηλανδία, παραδείγματος χάρη, όπου έχουν εγκαταληφθεί τα αποθέματα και δεν υπάρχουν επιδοτήσεις του Σαλής και Ισλανδία, όπως τα ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα με τις ε, διαπραγματεύσεις για τις παραχωρήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι αυτοί δεν θέλουν να μπουν ε, σε αυτό το σύστημα χορήγησης επιδοτήσεων αλλή. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό είναι καλό για τους ίδιου, αλλά πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλίας είναι να εφαρμόζει την κοινή ελεκτική πολιτική με βιώσιμο τρόπο. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που με στενοχωρεί ελαφρώς είναι η ερμηνεία της μείωσης διοξιδίου του άνθρακα. Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει ε, σε όλους τους κανονισμούς ε, με βάση τη στρατηγική του 2020 που καλούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά αυτό στην αλληλεία μπορεί να γίνει μόνο εφόσον αντικατασταθούν οι κινητήρες. Αυτή είναι η ερμηνεία που προσφέρεται, αλλά είναι λάθος. Η τροπολογία δική μας, η 1385, αναφέρεται σε αληπτικές μεθόδους λιγότερο ε, με μικρότερη κατανάλωση διοξιδίου του άνθρακα. Άρα δηλαδή, εάν τελικά χρησιμοποιούνται αυτές οι τράτες, ε, καταλαβαίνετε ότι ε, καταναλώνεται πολύ μεγαλύτερη ενέργεια από ότι αν χρησιμοποιούνται τα ε, παραδοσιακά εργαλεία. Αυτό που μας, επίσης μας ενδιαφέρει είναι η οικότοποι. Εκεί μπορεί να αποθηκευτεί, να δεσμευτεί το διοξίδιο του άνθρακα με την ε, βιώσιμη διαχείριση των ε, παράκτιων υδροβιότοπων. Τώρα, πιο κάτω, εκεί που γίνεται λόγος ε, για, τους, για τις περιοχές ανάκτησης της αλίας. Συμφωνήσαμε από αυτού στην έκθεση Ρόντες και εκεί πρέπει να δοθούν κονδύλια και νομίζω και αυτό θα συμβάλλει στην μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή θα υπάρχουν αλίες, ε, περιοχές χωρίς αλεία και εκεί θα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα. Μία άλλη τροπολογία που δεν την περάσαμε δυστυχώς στην έκθεση Ρόντες ήταν η τροπολογία μας σχετικά με τη μείωση των ενδυτικών επιπτώσεων ε, σχετικά με τη διαβίωση των ε, ζώων, αλληλευτικές δραστηριότητες και επιπτώσεις τους ε, στην διαβίωση των ζώων. Υπάρχουν κάποια προγράμματα για να αναπτυχθούν αλληλευτικές μέθοδοι οι οποίες δεν θα προκαλούν την ίδια ζημιά στη διαβίωση των ζώων. Αναφέρομαι ε, στα παρεπίπτοντα αλλιεύματα, ε, στα θηλαστικά, όλα αυτά που μπορούν να στηρίξουν ε, όλες οι ομάδες. Αναφέρομαι στις τροπολογίες 608 ε, και 1208. Τώρα, η τροπολογία μας 775 λέει ότι δεν θα πρέπει να δίδονται επενδύσεις ή μάλλον επιχορηγήσεις σε εκείνους τους τομείς όπου τα κράτη-μέλη δεν έχουν αποδείξει ότι υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην αλληλευτική ικανότητα και τους υπάρχοντες πόρους. Δηλαδή δεν θα πρέπει να δίδουμε τα χρήματα των ε, φορολογουμένων για την επιλεξιμότητα ή οτιδήποτε άλλο, εφόσον δεν γνωρίζουμε ότι η ικανότητα είναι σε ισορροπία με τους πόρους, γιατί αλλιώς κάνουμε επενδύσεις και μετά, αφού θα έχουν γίνει επενδύσεις, κοιτάμε να δούμε πώς θα ξεφορτωθούμε τα αλληλεπτικά σκάφη αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει πλέον να πάυσει να ισχύει. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν. Ευχαριστώ κύριε Τόμας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Από όσο το κατάλαβα θα πρέπει να πούμε μόνο τα κυριότερα θέματα. Πέντε παρατηρήσεις λοιπόν. Θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η Ο στόχο αυτού του ταμείου και η φιλοδοξία του είναι να γίνει μία αηφόρο δραστηριότητα, η αλληλευτική δραστηριότητα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει κάποιο λάθος στη μετάφραση της δική μου 307, fuel efficiency λέει, ενώ εγώ θέλω να πω energy efficiency. Κύριε Σιγητά, πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία μπορούμε σύντομα να συμφωνήσουμε, κυρίως για θέματα που αφορά την αύξηση των ελέγχων και την συλλογή των δεδομένων που είναι αποφασιστικής σημασίας. Κυρίως για το θέμα των δεδομένων, νομίζω ότι δεν θα πρέπει ο κανόνας που θα εφαρμόζεται να είναι η αρχή της προφύλαξης λόγω έλλειψης δεδομένων. Επίσης, συμφωνούμε με το θέμα της περιφερειοποίησης, ανάθεσης στις περιφέρειες κάποιων θεμάτων. Όπως έλεγε μία συνάδελφος, θα πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί, διότι πολλές φορές ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πιστεύω όμως ότι ο αρχηγός των τροπολογιών καταδεικνύει ότι μάλλον σε προσέγγιση απόψε αν θα φτάσουμε. Έγινε μια πρώτη συζήτηση τα θέματα της ε, ε, Διαφοροποίηση. Συμφωνώ. Αυτά που είπε και ο εισηγητή και πολλέ τροπολογίε που κατέθεσαν οι συνάδελφοι. Υπάρχει θέμα ορισμού μεταξύ ε, πολυδυναμικότητας και διαφοροποίησης. Νομίζω ότι η πολυδυναμικότητα θα πρέπει να λυθεί υπόψη δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη και το θέμα της διατροφής. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η ΚΑΛΠ είναι το μικρό κοριτσάκι της ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά θα δούμε δυστυχώς να αυξάνονται οι εισαγωγές αλλιευτικών ε, προϊόντων από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα συζήτησης που νομίζω ότι είναι σημαντικό είναι αυτό το οποίο αφορά τις ενισχύσεις για τα λιμάνια μετά την ε, ψηφοφορία που έγινε στο Στρασβούργο, δεδομένου ότι υποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι υποχρεωτική η εκφόρτωση των απορρίψεων, θα ήταν πραγματικά εκπληκτικό αυτό το κόστος να το επομισθούν οι τοπικές αρχές. Βεβαίως, οι τοπικές αρχές πρέπει να πω ότι είναι ε, αυτές που έχουν στη διάθεσή τους τα έργα υποδομή στα λιμάνια και θα πρέπει ό,τι γίνει να γίνει στα πλαίσια των κονδυλίων που θα δουν και στα πλαίσια του νέου αυτού ταμείου. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο θέμα της ανανέωσης του ολιευτικού στόλου και να πω ότι όλοι θα θέλαμε οι νέοι πραγματικά να ακολουθήσουν το επάγγελμα του αλλιέως. Και όλοι οι ευρωβουλευτές λένε ότι η ε, νεολαία είναι απόλυτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα πρέπει όμως τα λόγια να γίνουν έργα, βλέπουμε πολύ περισσότερους ενδιασμούς. Η συζήτηση ε, για αυτό το θέμα έγινε και από τον εισηγητή και από τους ε, συναδέλφους Ρόντους, Τρόμεβα και άλλους, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα στους νέους για να ακολουθήσουν αυτή τη δραστηριότητα με ελευτικό στόλο εκ 30 ετών. Με τραγικές πολλές φορές, με άθλιες συνθήκες, με δραματικές συνθήκες ασφάλειας. Υπάρχει στην Αλία ένα τριπλό αλφα. Εδώ έχουμε τριπλό α όπου έχουμε πάρα πολλά, τα περισσότερα ίσως επαγγελματικά ατυχήματα που οδηγούν σε ακροτηριασμού στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου έχουμε τους περισσότερες θανατηφόρους τραυματισμούς και παρά το γεγονό ότι κατανοώ αυτά τα οποία είπε ο κ. Στίβενσον για την ε, αποδοτικότητα, ναι, αλλά για να είναι κανείς αποδοτικός αλλιεύοντας, θα πρέπει να το κάνει στα πλαίσια μιας ισορροπίας. Συμφωνώ με το να αλλιεύουμε λιγότερο, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι εάν μειωθεί η ποσότητα θα πρέπει και η απόδοση να συνεχίσει να υπάρχει και για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να ανανεωθεί ο αλλιευτικός στόλος. Κυρίως για να μπορέσουμε να είμαστε ενεργειακά αποδοτικοί ώστε η επιλεκτικότητα να γίνεται σωστά και να δούμε πώς θα χειριστούμε τους πόρους που διαθέτουμε. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα πρέπει να υπάρχει ανανέωση του στόλου, λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά το θέμα της υπεραλίευσης. Δεν θέλουμε να υπάρξει αύξηση ελευτικής ικανότητας. Το είπε ορισμό, ο εισηγητής, αλλά το θέμα του ορισμού είναι σημαντικό. Οι υπηρεσίε του Κοινοβουλίου μα λέγουν ότι δεν υπάρχει ορισμό σε αυτό το θέμα. Όλοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την ελευτική ικανότητα και την υπεραλίευση. Το θέμα είναι εάν η ελευτική ικανότητα θα πρέπει να μετράται συνολικά, σφαιρικά, αλλά η η υπεραλίευση σε επίπεδο Ευρώπης θα πρέπει να γίνεται αναζώνη, αναλιευτική δραστηριότητα, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες ζώνες στις οποίες δεν υπάρχει αλλιευτική ε, υπερβολική ικανότητα και υπεραλίευση. Πώς μπορούμε λοιπόν όλα να τα βάζουμε στο ίδιο πακέτο για να βγάζουμε μέσους όρους. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ε, λεπτομεριακά και αναπερίπτωση ποια είναι η αλλιευτική ικανότητα και η υπεραλίευση χωρίς να τα βάζουμε, επαναλαμβάνω όλα, στο ίδιο σάκο και να βγάζουμε λάθος συμπεράσματα. Σταματώντας για τη μακρηγόρηση θέλω να πω ότι εγώ κατέθεσα τροπολογίες για να είναι χρονικά αηφόρος η αλλιευτική δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ώστε να μπορούν οι επαγγελματίες του κλάδου του που καταβάλουν προσπάθειες όσον αφορά την επιλεκτικότητα, την ε, ενεργειακή απόδοση και τη μείωση του διοξιδίου του άνθρωπη, που κάνουν ότι μπορούν ώστε να υπάρχει ασφάλεια επί των σκαφών κτλ. κτλ να έχουν ε, κάποια ενίσχυση από το Ταμείο το ευρωπαϊκό αυτό σε σχέση με τους υπολείπους που δεν τα σέβονται. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε κυρία Τόμας. Τελικά, ο κύριος Γκάλαχερ ζητάει το λόγο. I've come in a little bit late, so I'm not going to dwell on a lot of the uh, issues that were uh, raised previously, but suffice it to say that... Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι η δική μας η ομάδα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, στηρίζουν το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν δεδομένα που να αφορούν το μάρκετινγκ, της απορρίψης. Ε, κοιτάξτε, το θέμα είναι το εξής. Βεβαίως και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πρέπει να περιορίζονται οι απορρίψεις και για να γίνει αυτό ε, πρέπει να προσφέρουμε κίνητρα μικρής και μεγάλης κλίμακας στους ε, αλείς έτσι ώστε να αλλάζουν τα δίχτυα τους και ε, να έχουν διαφορετικά μάτια έτσι ώστε τα μικρά ψάρια να μένουν στη θάλασσα. Ε, όσον αφορά τώρα τα μικρά λιμάνια και τα νησιά, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ε, ριζοσπαστικοί με την εξής έννοια. Ε, στο τέλος ας μην ξεχνάμε ότι η έκθεση είναι δική μας και γι' αυτό ζητάμε από τον εισηγητή να εξετάσει τα πολύ μικρά λιμάνια και αυτό ως αποτέλεσμα των περικοπών θα διαπιστώσει μόνος του ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Νομίζω είναι σαφές ότι η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών επιθυμούν να εξεταστούν οι παράκτιες κοινότητες και τα λιμάνια. Η υποδομή έχει επιδεινωθεί, όπως είπα, δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Και μιλάμε για μικρές επενδύσεις, έτσι ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις σε αυτά τα λιμάνια και τα λιμάνια αυτά να ε, βελτιωθούν. Πρέπει λοιπόν ε, να προσφέρουμε και κάποια κονδύλια έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργείται πάγος, ε, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας πάγου στα λιμάνια, έτσι ώστε τα σκάφη που φτάνουν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον πάγο και δεν αρκεί να λέμε ότι δεν έχουμε πολλά λεφτά. Πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας αλλού. Η πλειοψηφία των αλλιέων βρίσκονται σε μικρά λιμάνια, ε, σε παράκτιες μικρές ε, κοινότητες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε τον προπολισμό της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εκεί ε, χρηματοδοτούν προγράμματα leader, που βοηθούν τις ε, μικρές ε, κοινότητες. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Βεβαίως ε, και εμείς μπορούμε να έχουμε κατά νου ότι το ταμείο αυτό χρηματοδοτεί κατά 45% και το υπόλοιπο πρέπει να χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις. Μιλάω πάντα για την χρηματοδότηση των μικρών λιμανιών. Και μιλάμε συνεχώς για τα, τις ποσότητες ε, ψαριών που έρχονται από τρίτες χώρες. Εδώ για μας υπάρχουν χρυσές ευκαιρίες και ξέρετε πώς μπορεί να γίνει αυτό με τις υδατοκαλλιέργειες. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε την Κομισιόν για την καθυστέρηση. Όλες οι χώρες ε, καθυστερούν γιατί υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσφέρεται χρηματοδότηση. Το επόμενο θέμα. ο στοχευμένος παροπλισμός. Ο παροπλισμός δεν είναι αγαπημένη λέξη, αλλά πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση. Να μάθουμε από το παρελθόν. Γιατί κατά το παρελθόν δόθηκαν χρήματα για παροπλισμό και αυτό ήταν απόλυτη διασπάθηση κονδυλίων. Τα σκάφη τα οποία παρέμειναν και παραμένουν θα πρέπει να είναι περισσότερο βιώσιμα. Ελπίζω λοιπόν ότι σε τελική ανάλυση ε, θα γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις, έστω και σε περιορισμένο βαθμό. Τελειώσαμε με τους ευρωβουλευτές. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πένας, εκ μέρους της Κομισιόν και μετά στον κύριο Κάντεκ. Χαιρόμαστε για τον πλούτο των σχολείων και των ιδιών που ακούστηκαν. Ευχόμαστε καλή τύχη και κουράγιο στον εισηγητή. Είναι τεράστιος ο αριθμός των τροπολογιών. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που μου ετέθησαν. Θα περιοριστώ, αν θέλετε, στο να σας εξηγήσω τη φιλοσοφία και τις αρχές ε, στις οποίες ε, βασίστηκε η Κομισιόν και θα αξιολογήσει μάλιστα και τις ε, προτάσεις τροπολογιών που συζητούμε. Βασική αρχή πιστεύω είναι ότι αυτό το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας, όπως και όλα τα διευθυντικά ταμεία που έχει προτείνει η Κομισιόν, είναι ταμείο που έχει ως ε, στόχο να εφαρμόσει την στρατηγική Ευρώπη 2020. Δηλαδή είναι όλα αυτά ταμεία ε, που θα προωθήσουν τις αλλαγές, αλλά δεν είναι ταμεία που θα διατηρήσουν το status quo δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα ήταν μη βιώσιμο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Οπότε ποιε είναι αυτές οι απαραίτητες αλλαγές. Ε, δεν μπορούμε βέβαια να προδικάσουμε την πολιτική διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο της εξέτασης του βασικού κανονισμού. Όμως, ε, ήδη έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένες ε, προτεραιότητες που ανεξαρτήτως των τελικών λεπτομεριών μας βρίσκουν όλους σύμφωνους. Όλοι συμφωνούμε νομίζω με την ιδέα ότι θα πρέπει η αλληλεία να οδηγηθεί προς, τα, προς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Όλοι συμφωνούμε ότι οι απορρίψεις είναι πρόβλημα που πρέπει να επιληθεί. Όλοι συμφωνούμε ότι εξαρτώμαστε υπερβολικά από τις εισαγωγές αλλιευμάτων και ενδεχομένω η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει μια λύση για τη μετρίαση αυτού της εξάρτησης. Όλοι ε, συμφωνούμε ότι ε, υπάρχουν ε, παράκτιες ζώνες που εξαρτώνται από την πέσκα, από την αλία, αλλά θα έπρεπε να εξαρτώνται και από άλλους οικονομικούς τομείς, από άλλες δραστηριότητες και όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε επαρκή διακυβέρνηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής με επαρκή χρηματοδότηση, επαρκή επιστημονικά στοιχεία κλπ. Σε όλα αυτά συμφωνούμε όλοι, είναι προτεραιότητές μας. Η οπτική της ε, Κομισιόν είναι ότι όσο περισσότερο συμπεριλάβουμε σε αυτόν τον κανονισμό άλλου τύπου μέτρα, τόσο λιγότερα χρήματα θα έχουμε για να επιτύχουμε τις πραγματικές μας προτεραιότητες. Ε, γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν πιστεύει ότι είναι σημαντικό ε, το Ταμείο όχι μόνο να περιοριστεί σε αυτές τις προτεραιότητες, αλλά να μην εστιάσει σε δύο συγκεκριμένες σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Τι δεν θα πρέπει να κάνει το Ταμείο. Πρώτον, να επαναλάβει λάθη του παρελθόντος. Και δεύτερον, να προσπαθήσει να διατηρήσει τέχνητα με δημόσια κονδύλια μη βιώσιμες ε, δραστηριότητες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα μικρό ταμείο όπως αυτό. Είναι σημαντικό να εστιάσει στις προτεραιότητές του. Α, ε, ορισμένοι οι βουλευτές μίλησαν για παράδειγμα και είπαν να συμπεριλάβουμε παρεμβάσεις για ε, ε, λιμενικές υποδομές, μεταποίηση κλπ. Συμφωνούμε ότι αυτές οι επενδύσεις είναι σημαντικές, είναι πολύ σημαντικές. Αλλά αυτές οι επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν και με άλλα ταμεία. Για παράδειγμα, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Γιατί εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα λίγα χρήματα τα οποία θα διαθέτει το Ταμείο μας για να χρηματοδοτήσουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ταμεία πολύ πιο ε, μεγάλα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εστιάσουμε, να συγκεντρώσουμε την προσπάθειά μας τις πραγματικές μας προτεραιότητες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Καντέκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πήραν το λόγο όλοι. Άκουσα όλες τις παρατηρήσεις. Που παρουσίασαν τι τροπολογίε που έχουν υποβάλει. Μια παρατήρηση για τον Ερνέστο Πένια, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ας σταματήσουμε, Σα αφορά πρόεδρε, ας σταματήσουμε να λέμε, να μιλάμε για μικρή επιτροπή, μικρό προπολογισμό, μικρό, μικρό, μικρό, όταν μιλούμε για την αλία. Ε, το έχω βαρεθεί αυτό. Προφανώς υπάρχουν ε, μεγαλύτερες επιτροπές, αλλά δεν είναι απαραίτητα νομοθετικές. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε και το λέω, δεν το λέω για εσάς, έτσι. Ε, δίνω, ε, προεκτείνω αυτά που είπες, ε, Γιατί μερικοί συνάδελφοι μας αποκαλούν μικρούς, μικρό το ένα, μικρό το άλλο. Μικρός προπολογισμό, μικρή επιτροπή. Εν πάση Δεν βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο μήκο σχήματο. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να συγκλίνουμε. Υπό ένα όρο. Υπό τον όρο. Ραούλ, άκουμε για να καταλάβεις. Με ένα όρο λέω. Να ε, συμφωνήσουμε επί της βασικής ιδεολογίας μας. Ε, κυρία Φράγα, εκτός μικροφώνου. Ε, δεν υπερβάλλω. Εσείς είσαστε ευρωβουλευτές, δουλεύετε. Γι' αυτό το λέω. Δεν θα πρέπει εντός αυτής της Επιτροπής να φέρουμε σε αντιπαράθεση, αυτό που θα επιθυμούσαμε να αντιπαρατίθενται μάλλον αυτοί που θα ήθελαν να διαλυθεί ο τομέα τη Αλία με αυτού που θέλουν να το διατρίσουν. Δεν πρέπει να αντιπαρατίθεται το Βορρά με τον Νότο. Δεν θα πρέπει να αντιπαρατίθεται τη θέμεθα ε, μεταξύ της ε, χρησιμότητας της ε, κρατικής παρέμβασης και της βλάβης που προέρχεται από αυτήν. Μεταξύ των πιο παρεμβατικών και των λιγότερο παρεμβατικών. Δεν θα πρέπει δηλαδή να μεταφέρουμε ιδεολογικές μάχες σε αυτή την Επιτροπή. Θέλουμε ένα ευρωπαϊκό βιώσιμο μοντέλο αλίας. Όλοι το θέλουμε αυτό. Αυτό είναι ο κοινό παρανομαστή. Στι συναντήσει μα με του κοινού ηγητές και με του ε, βουλευτέ, θα προσπαθήσουμε. Βλέπετε, έχουμε ένα ολόκληρο πάκο από τροπολογίε, Καταρχήν θα δουλέψω εγώ με του βοηθού μου για να υποβάλουμε προτάσει συμβιβασμού. Θα είμαστε επικοδομητικοί, με ανοιχτό πνεύμα, δεκτικοί και ελπίζω ότι όλοι θα καταφέρουν να δεχτούν το τελικό κείμενο έτσι ώστε η έκθεση αυτή να είναι πραγματικά παραδειγματική στο τέλος. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Muy bien, gracias, señor Πολύ καλά, ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Τώρα ας τα μανίκια μας και δουλέψουμε. Παίρνουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης 17. Δημιουργία κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλληψης της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Ήδη έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον προηγούμενο Νοέμβριο και σήμερα ο εισηγητής, ο κύριος Ρόμεβα, αυτό που θα κάνει είναι να παρουσιάσει το σχέδιο εκθεσής του. Του δίδω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα και την πρώτη φορά, έχουμε μπροστά μας βασικά μια έκθεση που αφορά την ε, λισαβονοποίηση. Δηλαδή, θέμα τεχνικο-νομικού περιεχομένου. Θέλησα λοιπόν εγώ από νομοθετικής πλευράς να κάνω κάτι πολύ απλό. Μία τροπολογία που έχει σχέση με το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τις πράξεις κατεξιδότησης σε σχέση με κάποιες παραγράφους και άρθρα και να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ίδια λογική που ακολουθήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις περίοδο τριετή κτλ. κτλ. Έκανα δηλαδή κάτι το οποίο είναι συνεκτικό με αυτό το οποίο ακολουθείτε εξαιτίας της εφαρμογής πολιτικής της Λισαβόνας και σε άλλες εκθέσεις. Τώρα, αυτό αφορά το νομοθετικό κομμάτι του θέματος. Το θέμα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι από πολιτική σημασία πάρα πολύ ευαίσθητο. Κυρίως μιλούμε για παράνομη αλληλεία και μηχανισμούς για να μπορέσουμε να ελέγξουμε αυτού του είδους την αλληλεία, την παράνομη λαθρεία και την άναρχη. Άρα, η συζήτηση είναι μια συζήτηση που γίνεται με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δεν είναι το τυχαίο ότι μετά από πολλά χρόνια, από πολλές παρεμβάσεις και πολλές αντιθέσεις, Πρόσφατα μας παρουσίασε η Κομισιόν τον κατάλογο των οκτώ κρατών που θεωρεί ότι δεν συνεισφέρουν και δεν συνεργάζονται ε, επαρκώς για να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τη λαθραλία και σήμερα, επαναλαμβάνω, έχει γίνει ένα πρώτο βήμα. Παραμένει όμως πρώτο βήμα, άρα επαρκές, Άρα είναι απαραίτητο και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε η Επιτροπή να εργαστεί πιο αποδοτικά ώστε να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία με το να συμπεριλάβει αυτές τις οκτώ χώρες που πρέπει να πω ότι δεν είναι οι κύριες χώρες που αφορούν την ποσότητα των λαθρέων αλλιευμάτων γενικά, αλλά ούτως ή άλλως να συμπεριλάβει και τις χώρες που πραγματικά όντως έχουν εξαιτία των ε, ε ικανότητα τους και της επιρροή τους συνεισφέρει πάρα πολύ σε αυτή την ε, άνερχη ελεία. Τη Φιλιππίνα, την Κορέα, και άλλες χώρες θέλω να αναφέρω. Και ας τολμήσουμε κάποια φορά να αναφέρουμε και την Κίνα που είναι μεγάλη απούσα από όλες αυτές τις συζητήσεις. Ας το θέσουμε επιτάπητο στο θέμα λοιπόν της Κίνας. Επιμένω, πρόκειται για ένα πρώτο κατάλογο για μια κίτρινη κάρτα, ούτε καν κόκκινη κάρτα. Για μια προειδοποίηση με κίτρινη κάρτα. Άρα πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Αλλά για τον λόγο αυτό, επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να υποφιληθούμε από τη δυνατότητα που μας δίδεται. Η συζήτηση αυτή περισσότερο από την έκθεση θα πρέπει όπως και ιδιωτικά να υπενθυμίσουμε την Κομισιόν ότι παίζονται εδώ πολλά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα το θέμα της αξιοπιστίας μας όσον αφορά την εξάλληση παράνομη λαθρέας και αναεξαλία. Και αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι και θέλουμε να απαιτήσουμε από άλλε χώρε να ενεργούν υπεύθυνα όταν ασκούν αυτή την δραστηριότητα, δεν θα πρέπει εμείς να έχουμε προϊόντα που δεν θα έχουν από κοινωνική και περιβαλλοντική πλευρά μια κάποια ε, εγγύηση. Και έτσι, για να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους την αλληλεία, θα πρέπει και τους πρωταθλητές να τους στοχοποιήσουμε. Αυτό είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η πιο σημαντική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, χώρες ε, τις οποίες ενοχλεί πάρα πολύ το ότι πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχουν χώρες που όταν πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον λένε ναι, αλλά όταν πρέπει να εφαρμοστούν τα κοινωνικά και οικονομικά μέτρα προβάλλουν ενδιασμούς. Ποια χώρα εννοώ? το Ηνωμένο Βασίλειο, ας το πούμε. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ σαφείς όταν αναφέρουμε ποιο είναι αυτό ο οποίο θέλει να βάλει τροχοπέδι σε τέτοιου βελτιώδεις. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι το θέμα αυτό και η συζήτηση επί αυτού του θέματος είναι πιο σημαντική από ό,τι γραφεί στην έκθεση. Θα ήθελα να επωφεληθώ από την παρουσία του κυρίου Πένιας για να κάνω και πάλι έκκληση όχι μόνο ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κρατών που θα συμπεριληφθούν στη λίστα αυτή, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε και μία λίστα των ε, σκαφών που πιστεύουμε ότι είναι κάπως συνένοχοι σε όλη αυτή τη διαδικασία της ε, άναρχης λαθρέας και παράνομης αλίας. Τελειώντα, θα πρέπει να πω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται αυτή τη στιγμή μία μελέτη. Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Δεν ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά ξέρω ότι κάποια στιγμή θα δούμε ποια είναι τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής που αφορούν εν μέρη τις ε, εισαγωγές αλλιευμάτων που προέρχονται από τέτοιες παράνομες αλλιευτικές δραστηριότητες. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ο σχετικός κανονισμός αυτός να είναι ένας από τους κύριους πυλώνες πρόσφυσης τη ΚΑΛΠ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ότι θα πρέπει στην εκπόνηση έκθεση αυτή να έχουμε συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι η κυρία πρόκληση εδώ δεν είναι να κάνουμε τον κανονισμό, αλλά να τον κάνουμε αποτελεσματικό και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το μέσο που θα δημιουργήσουμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτής της μελέτης να δούμε ποιες είναι, ποιοι είναι οι στόχοι του κανονισμού αυτή και βεβαίως ποιες είναι και οι κύριοι, ε, ε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι κυρίως ε, αντίθετοι σε αυτό και να μην αφήσουμε κάποιους να ε, κάνουν το σύστημα αυτό τέτοιο ώστε να είναι αναποτελεσματικό. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερος και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ η συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της μελέτης αυτής που θα ε, ολοκληρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το χρονοδιάγραμμα ίσως μπορούν πιο συγκεκριμένα να μας δώσουν ο Πρόεδρος ή η Γραμματεία. Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Πριν από κάποιες μέρες είχα θέσει κάποια ερωτήματα στον κύριο Ρόμβα και τώρα τα επαναλαμβάνω. Γιατί μου λέει ότι σε σχέση με την πρόταση Επιτροπής επιμένει στο 12.6 που αναφορά τα μικρά αλλιευτικά σκάφη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα θέματα της πιστοποίησης, νομίζω ότι στις ε, πράξεις εξουσιοδότησης θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι αντικείμενο, θα πρέπει να είναι το θέμα αυτό αντικείμενο συναπόφασης. Τώρα, Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει η Ισπανία. Μην πιστεύετε ότι το ζητάμε γιατί είμαστε κι εμεί από αυτού. Κάποια κράτη-μέλη ζητούν να υπάρξει αυτή η δυνατότητα. Θα ήθελα λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι το θέμα αυτό, ε, εάν ξέρουμε λεπτομεριακά περί τίνο πρόκειται, θα το προσέξουμε και θα το αφήσουμε στην εξοδότηση. Στο 16.1 αντιθέτω πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε. Ε, όχι κατ' εξουσιοδότηση πράξη, αλλά κατ' εκτέλεση. Νομίζω ότι αυτό αρκεί. Εκτελεστική. Επίσης, έχω σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τον κατάλογο των κρατών που δεν συνεργάζονται, 33.1. Κράτη λοιπόν που δεν συνεργάζονται. Εδώ έχω πολλές αμφιβολίες. Κατανοώ ότι πολλές φορές στη βιασύνη μας βάζουμε και βγάζουμε χώρες. Αλλά τώρα τελευταία, κύριε, βλέπουμε το θέμα των κρατών που δεν συνεργάζονται είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει μεγάλες αμφιβολίες το Κοινοβούλιο ότι η στάση της Επιτροπής είναι η πιο σωστή και την πιο κατάλληλη χρονική στιγμή. Πιστεύω ότι πολλές χώρες ούτε καν συμφωνούν με το να πρόκειται εδώ με πράξεις κατεξιοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ειλικρινά ότι σωστά το αφήνουμε σε αυτή την κατηγορία. Έχω μεγάλες αμφιβολίες όμως. Τώρα, αυτά ήταν τα κύρια θέματα που με απασχολώσουν. Επίσης εσείς Μιλήσατε για την εξουσιοδότηση κατά τη διάρκεια αυτής της τριετούς περίοδου. Κάνετε ένα σχετικό ερώτημα, αλλά θα ήθελα... Για το θέμα αυτό με το οποίο συμφωνούμε, την καταπολέμηση της παράνομης λαθρέας και ανεξελίας, να μου πείτε ότι αυτά τα οποία λέγει η Κομισιόν δεν αλλάζουν κατά πολύ το σύστημα. το Συμβούλιο ούτε καν το θεωρεί το θέμα αυτό ως θέμα ε, το οποίο μπορούμε να λύσουμε με τις πράξεις εξουσιοδότησης. Ε, λύστε μου την απορία μου, διότι πραγματικά πρέπει να σας πω ότι εγώ πραγματικά θέλω να προσέξω όλες τις λεπτομέρειες για να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε σωστά τα πράγματα. Σωστά τα πράγματα εμεί. Ε, τώρα, γιατί ξέρουμε τι γίνει και στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Φράγκα. Δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο, άρα δίδω το λόγο στην Κομισιόν πρώτα στον κύριο Πένια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ αυτά τα οποία είπε ο κύριο Ρωμέβα. Δηλαδή, ότι εκτό από τη συζήτηση αυτή τη εκτελεστική πράξη με στόχο να μην αλλάξει η πολιτική του κανονισμού, αλλά να τον προσαρμόσουμε στα πλαίσια της πολιτικής λισαβόνος. Αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου κάθε φορά που συζητούμε το θέμα αυτό πόσο σημαντικό είναι ο φάκελο αυτό. Είναι κάτι το οποίο πολλέ φορέ το επανέλαβα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί απολύτω τη σημασία που έχει το θέμα αυτό. Όπω όμω έχει ήδη, ή, όπως έχω ήδη αναφέρει, για να αιτιολογήσω γιατί αργούν οι διαδικασίε, είναι ότι δεν θα πρέπει εφαρμόζοντα τον κανονισμό αυτό να κάνουμε σφάλματα που θα διευκολύνουν περιπτώσεις στα δικαστήρια προσφυγής κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί αν δημιουργήσουμε προηγούμενο, εάν πάρουμε αποφάσεις βιαστικέ, εάν ε, δημιουργήσουμε μια κατάσταση που θα κάνει των πασών κάτι να προσφύγει εναντίον ημών στα ε, δικαστήρια, θα έχουμε καταστρέψει αυτό τον κανονισμό και για μας και για σας, αλλά περισσότερο για μας είναι πολλές φορές ε, απογοητευτικό το ότι υπάρχει τέτοια ε, αργοπορία σε αυτά τα θέματα. Αυτό όμως είναι απαραίτητο για να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρά ε, παρουσιασμένα επιχειρήματα για να έχουμε ένα σωστό φάκελο και να μην βιαστούμε. Διαφορετικά, όπως σας είπα, θα προσφύγουν κάποιοι εναντίον μας στα δικαστήρια και τότε ξέρουμε ότι η, η νομολογία όντα αρνητική θα μας οδηγήσει σε πλήρη καταστροφή. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Φράγκα, το 16.1 για μας είναι κατά κάποιο τρόπο μία τροπολογία της βασικής πράξης. Δηλαδή, έχει κάποιο νομοθετικό χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θα πρέπει να είναι πράξη κατεξουσιοδότηση. Αντιθέτως, στο άρθρο 33 είμαστε αποκλειστικά στην σφαίρα της εκτέλεσης. Εκτέλεση τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα νέο στοιχείο στον κανονισμό και κανένα νέο στοιχείο ε, δεν εκτιμάται. Υπάρχει εκτέλεση. Άρα έχουμε πράξη εκτέλεξης. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ε, ικανοποιήσει και να πείσει την ε, κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Καταλαβαίνω την δυσκολία της ε, Κομισιόν να κάνει αυτή την έρευνα εκ των προτέρων έτσι ώστε ε, να μην, ε, βρεθεί να μην εκτεθεί αν υπάρξει προσφυγή. Γι' αυτό το λόγο έστειλα αυτό το γενικό μήνυμα στην Κομισιόν. Περισσότερη, περισσότερο προσωπικό, περισσότεροι πόροι για αυτό το πράγμα. Δεν το λέω σε εσά προσωπικά, προ την Κομισιόν το λέω. Είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Και προκειμένου ακριβώ για να μην συμβεί, προκειμένου να μην συμβεί αυτό, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μα εκ των προτέρων και να διαθέσουμε περισσότερο προσωπικό και κεφάλαια, κονδύλια. Σχετίζεται βέβαια και με τη συζήτηση που είχαμε πριν από λίγο ε, με την ευκαιρία της έκθεσης ΚΑΝΤΕΚ για το ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της αλίας συγκεκριμένα. Τώρα, για τα δύο θέματα που έθιξε η κυρία Φράγα. Ομολογώ ότι ο μοναδικός στόχος δικός μου ήταν η λειτουργικότητα. Να εξασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα. Δηλαδή πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που ορισμένα αυτά μέτρα είναι πολύ περίπλογα και πολύ, και πολύ πολιτικής φύσεως. Και ορισμένα θέματα πραγματικά έχουν πολιτικοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μπορούμε να αντιδρούμε γρήγορα. Εμείς ε, στο Κοινοβούλιο πολύ συχνά ε, δεν εξασφαλίζουμε την ταχύτητα που απαιτούν οι καταστάσεις. Αυτή ήταν Αυτός ήταν ο δικός μου γνώμονας. Τώρα, είναι αλήθεια βέβαια ότι δεν βιαζόμαστε ιδιαίτερα να υιοθετήσουμε αυτή την έκθεση, οπότε ας μου δώσετε μία ακόμα εβδομάδα για να εξετάσω τις ε, τροπολογίες και να απαντήσω και στα ερωτήματα της κυρίας Φράγκα. Αν δεν σας ε, δημιουργεί πρόβλημα, δώστε μου άλλη μια εβδομάδα. Αν είναι δυνατόν. Είναι ένα θέμα το οποίο ε, εύκολα θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με την κυρία Φράγα. Κυρία Φράγα θέλει το λόγο, όχι. Ωραία. Εγώ θα έλεγα να υποβληθούν τροπολογίες μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Αλλά πραγματικά δεν βιαζόμαστε. Οπότε αν θέλετε αναβάλουμε κατά μία εβδομάδα αυτή την ε, προθεσμία. Κανείς δεν έχει αντίρρηση. Με μικρόφωνο όμως παρακαλώ. Αν έχετε αντιρρήσεις. Ωραία. Ε, αναβάλουμε την ε, ε καταληκτική μορφή για την υποβολή τροπολογιών κατά μία εβδομάδα. Και μετά θα δούμε την ψηφοφορία της ε, στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Περνάμε στο σημείο 7. Τροποποίηση του κανονισμού 1100 του Συμβουλίου. Ανάκτηση των, του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χελιών. Θα θυμάστε ότι τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο, η Κομισιόν μας έκανε την παρουσίαση του κανονισμού και τον Ιανουάριο ανταλλάξαμε τις πρώτες, ε, για πρώτη φορά απόψεις ε, για αυτή την πρόταση. Η συγγήτρια η κυρία Λοβίν. Σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης που έχει υποβάλει πλέον η κυρία Λοβίν. Έχετε το λόγο. Ε, thank you very Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ζητήσω ε, συγγνώμη από τους συναδέλφους γιατί υπάρχουν κάποια λάθη στην έκθεση. Ε, ένα λάθος που έγινε από τη γραμματεία. Η τελευταία εκδοχή της ε, έκθεσης δεν δόθηκε προς μετάφραση, αλλά η πρώτη τελευταία. Και εντοπίσαμε τουλάχιστον τρία σημεία όπου ε, δεν μας άρεσε το κείμενο. Θα επανέλθω, εν πάση περιπτώσει, αυτό. Αυτό το θέμα ήταν πολύ δύσκολο. Βεβαίως πρόκειται για λισαβονοποίηση, μια που σε αυτή τη διαδικασία. Από την άλλη, με τις ε, νέες ε, επιστημονικές, ε, τα νέα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τα αποθέματα χελιού, δεν είναι νέα πρέπει να πω, είναι δεδομένα που απλά επιβεβαιώνουν όλο και περισσότερο την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται το απόθεμα του χελιού. Άρα δηλαδή πρέπει να δούμε λιγάκι την κατάσταση εδώ και αρκετά χρόνια έχει αποδειχθεί ότι δεν λαμβάνονται υπόψη όλα τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν εντωμεταξύ προκύψει. Ήδη το 2007 το ευρωπαϊκό χέλη συμπεριλήφθηκε συμφωνία Τσίτες στο παράρτημα 2 όπου προβλεπόταν ότι θα πρέπει ε, να μην υπάρχει εμπόριο αυτού του είδους που απειλείται από αφανισμό. Αυτή η συμφωνία ΣΥΤΕΣ ε, πέρυσι για πρώτη φορά έκανε λόγο για ανασύσταση του αποθέματος. Ε, ο κανονισμός προβλέπει αυτό ως μέτρο στο οποίο μπορούν να καταφύγουν τα κράτη-μέλη για να επιτύχουν το στόχο του 40% ανασύσταση. Τώρα, οι ISIS ε, είναι πολύ προσεκτική σχετικά με αυτά τα μέτρα της ε, ανασύστοσης, ε, διότι δεν είναι σίγουροι ότι υπάρχουν πλέον πλεονάσματα στην Ευρώπη που να μπορούν να μεταφορτούν σε άλλες περιοχές. Αυτά λέει η ISIS, το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών. Επίσης, στα προγράμματα ανασύστασης ε, δεν προβλέπεται κανένα μέτρο που να αφορά στις συνθήκες με τις οποίες ε, ενδεχομένως μπορεί να γίνει ανασύσταση του αποθέματος. Έτσι λοιπόν, ορισμένα κρατημέλη κατέφυγαν ε, σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το μέτρο, αλλά πάλι άρχισαν σιγά σιγά να το χρησιμοποιούν δειλά, μόλις τέθηκε σε ισχύ. Ε, εν τω μεταξύ όμως πρέπει να πω ότι η αλληλεία χελιού έκτοτε έχει αυξηθεί και γι' αυτό λοιπόν ε, εκείνο που δεν μπορώ να παραδεχτώ είναι τα στοιχεία εμπορίου. Ένα κιλό, όπως ξέρετε, θα μπορούσε να πουλτεί 600 ή 700 ευρώ. Και από τότε που προέκυψε ο κατάλογος CITES το 2009, απαγορεύεται το διεθνές εμπόριο χελιού, γιατί είναι ένα είδος που απειλείται θανάσιμα από αφανισμό. Εκείνο όμως που ανακαλύψαμε κατά τη διαδικασία σύνταξης της έκθεσης είναι ότι τα στοιχεία εμπορίου αυτού του είδους δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία αλίας που σημαίνει ότι τουλάχιστον δύο κρατή, η Γαλλία και η Ισπανία, έχουν μεγάλες ε, ποσότητες ε, χελιού, αλλιεύουν χέλ και δεν το καταγράφουν. 15,7 τόνους χελιού που δεν καταγράφεται. Αυτό ισχύει τώρα. Μιλάμε για 15.700 κιλά, χελιού με περίπου εκτιμόμενη αξία 11 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για εμπόριο, παράνομο εμπόριο γόνων ενός ε, είδους που απειλείται θανάσιμο από αφανισμό. Εκείνο που με απασχολεί πάρα πολύ σε σχέση με το πρόγραμμα ανασύστασης αποθεμάτων είναι ότι δεν προβλέπονται προϋποθέσεις για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανασύσταση. Και το μέτρο αυτό θα έλεγα ότι υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ως προκάλημα ή μάλλον για τη συγκάλυψη Παράνομο εμπορίου χελιού, δηλαδή ε, θα πολλούνται οι γόνοι χελιού στην ασιατική αγορά με πολύ μεγάλο κέρδος. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και το απόθεμα που θα έπρεπε ίσως να σταλεί στην Βαλτική θάλασσα ή αλλού, έτσι ώστε να υπάρξει ανασύσταση του αποθέματος του ευρωπαϊκού χελιού και αυτό είναι πολύ αμφίβολο. Έτσι λοιπόν ε, το ε, Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας, ΆΙΣΕΣ, λέει ότι ε, καταρχήν δεν είναι σίγουρο τι θα γίνει με το γόνο, διότι μεταφέρεται αλλού και δεν είναι σίγουρο πώς θα καταλήξει. Μετά επειδή είναι μακριά οι αποστάσεις και καταναλώνουν το λίπος τους, δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν ε, στον προορισμό. Ε, κατόπιν, το Διεθνές Αυτό Συμβούλιο λέει ότι ε, μπορούν να μεταφερθούν με τα μέτρα ανασύστασης και οι ασθένειες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και προειδοποιήσεις ε, από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών σχετικά με αυτό το μέτρο ανασύστασης αποθεμάτων. Έτσι λοιπόν ζητάμε από την Κομισιόν να αξιολογήσει το εμπόριο χελιού και επίσης και να λάβει υπόψη της ε, τις ε, συμβουλές ε, του Διεθνού Συμβουλίου για την ανασύσταση αποθεμάτων και αυτές τις συμβουλές να τις εντάξει στα προγράμματα που θα εκπονήσει. Τώρα, αν δούμε λιγάκι την έκθεση, θα διαπιστώσουμε το εξής. Προσπαθήσαμε να μην μπούμε στον στόχο. Ο στόχος είναι το 40% αυτών των χελιών θα μπορούσαν να έχουν ε, καταφύγει στη θάλασσα του Σαργκάσο. Αυτό ε, ποτέ δεν το αξιολόγησε το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών. Ίσως να μην είναι και ικανοποιητικό ο στόχος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν το θίξαμε αυτό. Πολλά πράγματα προσπαθήσαμε να μην θίξουμε, αλλά προσθέσαμε εδάφια που νομίζω ότι τοποθετούν το πλαίσιο του όλου θέματος. Η τροπολογία 1 αναφέρεται στο παράρτημα της σύμβασης ΣΑΙΤΕΣ. Η δεύτερη τροπολογία αναφέρει ότι από το 2010 τα ευρωπαϊκά χέλια βρίσκονται στο κατάλογο όσοι απειλούμενα είδη. Τροπολογία 3 λέει ότι βλέπουμε τις τελευταίες συστάσεις του Διεθνούς Αυτοσυμβουλίου του ISIS που επίσης ε, συστήνει η ε, αλληλεία και άλλες ανθρώπινες ε, δραστηριότητες που απειλούν τα χέλια να περιστούν ή δυνατόν κοντά στο μηδέν, να μηδενιστούν. Ε, και αν δεν έχετε αυτή την εκδοχή μπροστά σας θα σας δώσουμε αργότερα την τροπολογία. Επίσης ε, προσθέτουμε ένα εδάφιο που αναφέρει τι λέει το Διεθνές Συμβούλιο για το πρόγραμμα ε, που λέει ότι δεν μπορεί το, να ανασυνταχθεί ουσιαστικά ο πληθυσμός των χελιών. Στην τροπολογία υπαριθμών 5 έχουμε το αρχικό κείμενο. Εκεί γίνεται λόγος ε, για χέλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανασύσταση, βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν κάποιες ε, προδιαγραφές και ότι πράγματι η αύξηση του πληθυσμού θα οδηγήσει σε ανασύσταση του στόχου. Κατόπιν, κάναμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή διαγράψαμε ένα άρθρο το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο και υπήρχε στον κανονισμό. Πρόκειται για την ε, αξιολόγηση των τιμών της αγοράς. Προβέπεται λοιπόν ότι αν μειωθεί η τιμή του χελιού, σε σχέση με τις τιμές ε, χελιού που χρησιμοποιούνται για άλλα μέτρα, θα πρέπει να υπάρχει ε, προσωρινή μείωση των χελιών που χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό του αποθέματος. Άρα δηλαδή το 60% των ε, χελιών που ψαρεύονται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό του αποθέματος. Το άρθρο όμως αυτό λέει ότι αν υπάρχει αν διαφορά μέσα στην τιμή των χιλιών που χρησιμοποιούνται για τον εμπλισμό του αποθέματος με ε, τα άλλα χέρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για άλλους σκοπούς, μπορεί ο στόχος να περιοριστεί κατά 60%. Αυτό λοιπόν το άρθρο ε, μέχρι τώρα δεν το σεβάστηκαν τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη μέχρι το 2011 έπρεπε να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Κομισιόν για την αξιολόγηση των τιμών της αγοράς. Και δεν έγινε αυτό. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν στην πρόταση της λισαβονοποίησης ε, το 2011 το μετέθεσε στο 2013, έκανε ήδη δηλαδή αυτή την αλλαγή και νομίζω ότι το, αυτό το άρθρο πλέον είναι παντελώς απαρχαιωμένο ε, και αντιπαραγωγικό, πλήρω αντιπαραγωγικό. Δεν νομίζω ότι ε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Και εν πάση περιπτώσει η Κομισιόν θα προτείνει, θα καταθέσει νέα πρόταση και νέο κανονισμό. Αυτό λοιπόν τώρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να δούμε λιγάκι τα στοιχεία περί εμπορίου. Εμείς αυτό προτείνουμε. Τροπολογία 10. Τη διαγράφουμε σχετικά με τη μείωση των μέσων τιμών αγοράς. Αυτή έχει σχέση και με την τροπολογία 11 και 12 και εδώ προτείνουμε τη διαγραφή γιατί είναι η ίδια διάταξη που αφορά στην αξιολόγηση των τιμών της αγοράς. Κατόπιν δυστυχώς έχει παρισφρήσει ένα λάθος. Τροπολογία υπερτιμών 13. Εδώ λέει ότι το άρθρο 3 απαλήφεται, αλλά δυστυχώς δεν θα έπρεπε να λέει 3. Είναι το άρθρο 2 που ε, απαλήφεται και πιο κάτω λέει αντικαθίσεται. Αυτό, με πάση δημιουργεί κάποια σύγχυση. Επίσης, για τα πρακτικά να καταγραφεί δεν πρόκειται για μεγάλη αλλαγή, αλλά στην τροπολογία υπερθμών 14 έχουμε προσθέσει σε ένα από τα μέτρα θα μπορούσε να είναι η μείωση και αν είναι αναγκαίο η απαγόρευση της εμπορικής ελληνικής δραστηριότητας. Προσθέσαμε δηλαδή την απαγόρευση. Και αυτό δεν αλλάζει την ουσία, γιατί έτσι και αλλιώ αυτό μπορούν να το κάνουν τα κράτη-μέλη και ένα κρατος μέλος έχει ήδη καταφύγει σε αυτό το μέτρο. Η Ιρλανδία έχει ε, επιβάλει την απαγόρευση της ε, αληφτικής, εμπορικής αληφτικής δραστηριότητας. Και η τροπολογία υπερθών 16 και αυτή ε, μπορεί να διευκρινίσει, ή ο στόχος είναι να διευκρινίσει την κατάσταση από το maybe πάμε στο shall στα αγγλικά η τροπολογία υπαρθμών 18 και αυτή προβλέπει τη διαγραφή της διατύπωσης ε, που λέει έλεγχος των τιμών της αγοράς. Τροπολογία 19 Πιστεύουμε ότι ο ρυθμός ε, αναφοράς από πλευράς ε, κρατών μελών δεν θα πρέπει να μειώνεται μετά την πρώτη έκθεση ε, τριετή έκθεση, ο ρυθμός να μην μειώνεται, αλλά τον αντίον να επιτείνεται. Να γίνονται δηλαδή εκθέσεις πιο συχνά, αυτό σημαίνει. Ίσως σε αιτήσια βάση και τα στοιχεία θα αποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, λαμβάνοντας υπόψη το πόσο επίγουσα είναι η κατάσταση ε, σχετικά με τα αποθέματα χελιού. Η τροπολογία 20 ίσως είναι πλέον επίμαχη. Και λέμε εδώ, ότι αν αυτό το Διεθνές Συμβούλιο το ISIS ε, επιβεβαιώσει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα αποθέματα, να ανασταλούν όλα τα μέτρα μέχρι να ε, τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός με βάση την πρόταση. Αυτά το αργότερο το 2014. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία που τρέχει, ότι η Κομισιόν περιμένει την αξιολόγηση των προγραμμάτων διαχείρισης ε, χελιού ε, σχετικά με την πρόοδο κυρίως που έχει επιτευχθεί, το Διεθνές Συμβούλιο ε, ISIS για την εξερεύνηση των θαλασσών, το Συμβούλιο αυτό επιλήφθηκε του θέματος και ακούσαμε ότι τα στοιχεία που υποβλήθηκαν μέχρι τώρα από τα κράτη-μέλη δεν επαρκούν, ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Αυτή η διαδικασία λοιπόν ε, τρέχει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρόβλημα με, το, με τα χέλια ξεκίνησε πριν από πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια όταν η Κομισιόν άρχισε να απευθύνεται στα κράτη-μέλη προσπαθώντας να τα πείσει να λάβουν μέτρα. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Τα κρατη ε, δεν επιθυμούσαν ε, να λάβουν μέτρα, ούτε και να καταθέσουν στοιχεία και το Διεθνές Συμβούλιο, ISIS, ε, επισήμενε και επισημαίνει συνεχώς το πρόβλημα με τα αποθέματα. Ίσως η κατάσταση το μεταξύ να έχει επιδεινωθεί και γι' αυτό πράγματι είναι πλέον επίγον να υπάρξει κάποια πάυση και να δούμε πότε και πώς μπορούμε να επιτρέψουμε και πάλι την αλία και να είμαστε σίγουροι όμως ότι αυτό δεν θα οδηγήσει στον ε, αφανισμό αυτού του επαπειλούμενου είδους και ευχαρίστω να ακούσω τις απόψεις σας, τις απόψεις των συναντέλφων επί του θέματος και προσβλέπω μεγάλη χαρά στη συνεργασία με όλους τους κοιόδης εισηγητές. Σας ευχαριστώ κυρία Λόβιν. Κυρία Φράγκα. Έχω αρκετά προβλήματα με την έκθεση. Πρώτα απ' όλα, είναι θέμα διαδικασίας. Στην επιτροπολογία Πιστεύω ότι πλην εξαιρέσεων και υπήρξαν εξαιρέσει, ακόμη και σε μία πρόταση Επιτροπής που ζητά να αλλάξει οι τιμές της αγοράς έτσι όπως προβλέπεται στον κανονισμό, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποφεληθούμε από μία πρόταση προσαρμογής της επιτροπολογίας για να αλλάξουμε ένα κανονισμό. Και αυτός ο κανονισμός το είδαμε και το ζήσαμε και είχαμε την εμπειρία, κανονισμό για τον οποίο γίνανε συζητήσεις σε έντονο πνεύμα. Και εδώ και στο Συμβούλιο μέχρι να καταλήξουν τη συμφωνία. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να κάνουμε αλλαγέ ε, έτσι όπως τις προτείνει ο κύριος Λέβιν. Συμφωνώ με κάποιε, αλλά με την αρχή δεν συμφωνώ. Επίση, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που δεν καταλαβαίνω. Η έξι τι καινούριο προσφέρει. Διότι ό,τι το λέει εδώ προβλέπεται στο άρθρο 7. Αυτή είναι η γενική παρατήρηση. Δεύτερον, δεν συμφωνώ επίσης να αλλάξει πλήρω η νομική βάση του 290. Πράξεις καταξιοδότης να γίνουν εκτελεστικές. Διότι νομίζω ότι η αρχική πρόβλεψη έχει γίνει σύμφωνα με τις αρχές αυτού του κανονισμού. Τώρα, αν κάποιο τους ε, ενδιαφέρει περισσότερο από άλλους να υπάρχουν πράξεις καταξιδότηση για να τις ελέγχουν καλύτερα, είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η αλλαγή να προβλεφθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και στα πλαίσια του 290 και 290 που είναι η νομική βάση, τι θέλετε να κάνετε, να μας αφαιρέσετε και αρμοδιότητες που έχουμε ώστε να ανακαλέσουμε μια κατάσταση. Άρα δεν συμφωνώ ούτε τύπης ούτε επί της ουσίας με αυτήν την έκθεση της κυρίας Λοβάν. Για κάποια θέματα επιμέρους θα μπορούσα να συμφωνήσω, αλλά επιμένω. Δεν ε, έχοντας ακούσει την παρουσίαση ότι δεν θα πρέπει να θα από τις ανθρώπες μας δίνει επιτροπή Πολλογία για να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεύτερον, δεν συμφωνώ από πράξει. Κατογιώ να περάσουμε σε εκτελεστικέ. Διότι εδώ δεν υπάρχει λόγο ε, ύπαρξη αυτή τη έκθεση. Αυτά θέλω να πω. Ο κύριο Κούν. herzlichen Dank an die Berichterstatterin. Ευχαριστώ πολύ την ε, εισηγήτρια και ευχαριστώ και την κυρία Φράγκα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να συζητήσουμε σε επίπεδο αρχής. Δηλαδή, οι κανονισμοί που προσαρμόζονται με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, πώς οι κανονισμοί αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν με τεχνικής φύσεως εργαλεία. Ε, εάν θέλουμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, πρέπει να το βάλουμε στη μερίσια διάταξη, γιατί τελείω τα μπερδεύουμε και τα συγχαίουμε. Ε, και η κυρία Φράγκα το είπε και εγώ το πιστεύω, ήδη το 2007 είχε προκύψει αυτό το πρόβλημα ότι το απόθεμα του Ευρωπαϊκού Χελιού αντιμετώπιζε προβλήματα, αντέδρασε η Κομισιόν και το Συμβούλιο και συζητήσανε ε, για το σχετικό κανονισμό. Τότε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό θέμα που είχε προκύψει ήταν ότι η αλία, η ε, πώληση ε, χελιών μικρών ή μεγάλων, χελιών που έτυχαν μεταποίησης ή όχι, αυτό απαγορεύτηκε πλήρως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να απαγορευτεί αυτή η πώληση των μικρών χελιών για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χέλια για την αναπαραγωγή. Αυτή ήταν η απόφαση που ελήφθη. Και έτσι λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη ήταν υποχρεωμένα να λάβουν μέτρα έτσι ώστε το ευρωπαϊκό χέλι να πολλαπλασιαστεί στις γνωστές οδούς που υπήρχαν και υπάρχουν. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Και έχουμε λοιπόν ε, το ε, Γενικό αυτό Διεθνές Συμβούλιο και πολλοί άλλοι που όμως ε, δεν μπορούν να αποφανθούν κατά πόσον τα μέτρα απέδωσαν ή όχι. Η διαπίστωση καταρχήν είναι ε, βέβαια ότι υπάρχει μια θετική τάση και αυτό το δέχονται όλοι οι επιστήμονες. Ε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δεχτούμε ή να θεωρήσουμε ότι τα χέλια θα έρθουν από τη θάλασσα των Σαργασών στις δικές μας τις ε, γνωστές θάλασσες. Πάντως όλοι λένε υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Όσον αφορά τώρα τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, και τον κανονισμό και όλα τα άλλα, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς ε, θα κάνουμε. Όμως ε, εγώ πιστεύω σε επίπεδο αρχής, ε, σας λέω, σας λέω, το να τα αφήσουμε όλα στα χέρια των επιστημόνων, είτε πρόκειται για τον κατάλογο ΣΥΤΕΣ, είτε για το ΙΣΕΣ, ε, το Διεθνές αυτό Συμβούλιο Εξερεύνησης των Θαλασσών, είτε πρόκειται για την καταγραφή σε καταλόγους, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις αρμοδιότητές μας ως Κοινοβούλιο, μαζί βέβαια με την Κομισιόν και το Συμβούλιο, και να μην ε, αντιδράσουμε υπερβολικά, διότι εξακολουθεί να είναι απαραίτητο τα προγράμματα εμπλουτισμού του αποθέματος ε, των χελιών, ε, τα προγράμματα αυτά να λειτουργήσουν. Βεβαίως και θα πρέπει κάποια χέλια να μεταφερθούν ε, σε οδούς προς τα πάνω, προς τη Βόρεια Θάλασσα, προς τη Βαλτική. Ε, θα πρέπει τα χέλια να μπορούν και να ζουν στις ε, εσωτερικές θάλασσες, αλλά από τη στιγμή που βρίσκονται σε ηλικία αναπαραγωγής να μπορούν να μεταφερθούν στο τρίγωνο των Βερμουδών στις θάλασσες των Σαργασών. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί αν αρχίσουμε να λέμε καθαρά δυνητικά, μα ενδέχεται τα αποτέματα να επιδεινωθούν, μα ενδέχεται οι επιστήμονες να μην γνωρίζουν και ας το αφήσουμε λιγάκι και θα δούμε και για ένα χρόνο ε, δεν θα επιτρέπεται η αλία, γενικά η αλία του χελιού είτε για μικρών είτε μεγάλων χελιών Αγαπητή κυρία Λεβίν, κοιτάξτε τώρα το να θέλετε να βάλετε τιμές αγοράς σε έναν κανονισμό που θέλουμε να προσαρμόσουμε με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό εγώ το βρίσκω προβληματικό. Εξάλλου, εγώ πιστεύω ότι ο κανονισμός που προτείνει η Κομισιόν από κοινού με τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να τεθεί απότομα εκτός ισχύς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρετε δεν έγινε τίποτα και πρέπει να λάβουμε ριζικά μέτρα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την απαραίτητη βάση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, γιατί εμείς επιθυμούμε τα αποθέματα σταδιακά να ανακάμψουν. Επιθυμούμε όμως το χέλι να υπάρχει για μας στην Ευρώπη, να προσφέρεται γιατί όχι, και στους αλληλείς ε, και γιατί όχι στο δικό μας τον οικότοπο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά πιστεύω ότι μια καλή πρόταση θα προκύψει μόνο εφόσον μπορέσουμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία. Θα είμαι σύντομος. πήρα μόλις σήμερα το κείμενο στη γλώσσα μου ε, και το διέτρεξα βέβαια. Ξανασυζητήσαμε το θέμα αυτό το Γενάρη και η συγγήτρια άκουσε τα σχόλιά μας. Καταρχήν να πω ότι η πολιτική μου ομάδα θα προτείνει να ε, καταγράψουμε πως ε, το χέλι βρίσκεται σε μια... Ε, διατρέχει κίνδυνο εξαφάνισης. Συνεπώς δεν πρέπει να περιοριστούμε στην λισαβονοποίηση του, του κειμένου. Βέβαια, έχουμε διαφορετικές ε, απόψεις για το πώς μπορεί να ανακτηθεί το απόθεμα των χελιών. Έχουμε κάποια επιστημονική γνώση, αλλά δεν είναι επαρκής. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Επίσης υπάρχει που πάνε πολύ ερωτηματικά για το ποιο θα λάβει ποιο ρόλο. Ορισμένα προγράμματα διαχείριση ε, δεν λειτουργούν σωστά, συνεπώ θα πρέπει να δούμε ε, διάφορα ζητήματα σε σχέση με αυτέ τι εκκρεμότητε. Επίση, το θέμα των πράξεων κατεξουδότηση και των εκτελεστικών πράξεων και ποια είναι καλύτερη. Ε, πάντως, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα πάντοτε ότι τα χέλια διατρέχουν τον κίνδυνο αφανισμού. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Muchas gracias. Bueno, ha finalizado la intervención de los diputados. Vamos a dar la palabra a la... Θα δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν, αφού τελείωσαν οι συνάδελφοι βουλευτέ, κ. Μπιάνκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν ε, θα θέλαμε να συγχαρούμε την κυρία Λεβίν ε, που κατέθεσε αυτήν την ε, πρόταση. Εμείς είπαμε ότι ε, δεν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με αυτό το θέμα γιατί βρίσκεται στη διαδικασία προσαρμογής ε, στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καταθέσαμε αυτή την πρόταση με τη μορφή που βλέπετε. Η κυρία Λεβίν έφτιαξε μία σειρά θεμάτων και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά την κατάσταση του αποθέματος χελιού, που πράγματι είναι προβληματική. Και αυτό φαίνεται και στην ετήσια έκθεση του ISIS, του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης των Θαλασσών. Όπως είπε και ο εισηγητής, προσπαθούμε τώρα να δούμε πώς λειτουργήσε ο κανονισμός. Εξετάσαμε τις πρόσφατες επιστημονικές ε, ή θα εξετάσουμε τις επιστημονικές προτάσεις κατά τον Ιούνιο-Ιούλιο εάν τα κράτη-μέλη μας δώσουν τις προτάσεις τους ε, έγκαιρα. Και όπως προβλέπετε στον κανονισμό προβλέπουμε να καταθέσουμε την πρότασή μας κατά το τέλος του έτους. Αυτός λοιπόν είναι ο προγραμματισμός ε, που είχαμε κάνει. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχουν πολλές ε, ανησυχίες, τις ακούσαμε αυτές σήμερα και έχουν ε, σχέση βεβαίως με όλα αυτά τα οποία κάνουμε εμείς. Εμείς ε, θα θέλαμε να μπορούμε να εντάξουμε στις προτάσεις που κατατέθηκαν και τις, τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου ISIS. E θα σας εξηγήσω λιγάκι πώς προέκυψε αυτή η πρόταση. Εμείς ήμασταν πολύ συγκρατημένοι, διότι όπως σας είπα ήμασταν στη διαδικασία προσαρμογής στη συνθήκη της Λισαβόνας και γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε να καταθέσουμε ε, μία έκθεση για τον κανονισμό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ό,τι και αν συμβεί, όποια κατεύθυνση και αν αποφασίσει να ακολουθήσει το Συμβούλιο, πολύ σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα να εξετάσουμε τις ανησυχίες της κυρίας Λόβιν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ε, κυρία Λόβιν. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Όσον αφορά τώρα την επιτροπολογία και τη διαδικασία προσαρμογής στη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, νομίζω ότι τα έχω σχολιάσει όλα αυτά και ε, θέλω να σας πω ότι δεν ήταν εύκολο για μένα να γνωρίσω ε, τη διαδικασία της επιτροπολογίας και προσαρμογής στη συνθήκη της Λισαβόνας. Βλέποντας όμως ε, το χρονοδιάγραμμα που διέτρεξε αυτός ο κανονισμός όλα αυτά τα χρόνια, ανησύχησα, σκέφτηκα ότι δεν θα γίνει τίποτα και πρέπει να καταθέσω αυτές τις προτάσεις. Τα κράτη-μέλη κατέθεσαν ε, πολυκαθυστερημένα τα προγραμματά τους, την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Ε, δεν υπήρχε καμία συνοχή στις ημερομηνίες ε, που κατέθεσαν και εγώ προέβλεπα ότι και η διαδικασία της αξιολόγησης θα ήταν ε, πολύ αργή και οι διαπραγματεύσεις, γιατί έβλεπα ότι όλα καθυστερούσαν, σέρνονταν, αν μου επιτρέπετε, και εντωμεταξύ αυτό που λέει το Διεθνές Συμβούλιο ε, είναι σαφές, σαφέστατο κάθε χρόνο, λέει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει σχεδόν καθόλου αλία ε, χελιού. Και εμείς κατ' ουσίαν το γνωρούμε αυτό. Για δέκατη συνεχή ε, χρονιά το λέει το Διεθνές Συμβούλιο απαγορεύστε την αλία χελιού. Κυρία Φράγκα, όσον αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι καλύτερο να υπάρχουν ε, από τις ε, εφαρμοστικές πράξεις. Αλλά στις ε, τροπολογίες 11 και 12... Αυτή είναι η μόνη πρόταση της Κομισιόν για κατεξοδότηση πράξης και λέει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις ε, κατατεξιδότηση πράξεις ε, για να ε, προβεί στην αξιολόγηση και τον έλεγχο. Δεν ξέρω αν ισχύει σήμερα το να δούμε τι θα κάνουμε με την ε, μείωση της τιμή του χελιού. δεν ισχύει όμω αυτό, αποφασίσαμε να τα διαγράψουμε. Διαγράφουμε την ε, τροπολογία 11 και 12 και όλες τις αναφορές στις κατεξουσιοδότηση πράξη. Κύριε Κούνε, Βέρνα, αγαπητέ Βέρνα, είπατε ότι απαγορεύτηκαν οι εξαγωγέ σωστό αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν δει κανεί τα στοιχεία αλίας, Ε, αλλιεύονται περισσότερα μικρά χέλια από αυτά που εμφανίζονται στην αγορά. Τείτε λοιπόν το εξή μεγάλο ερώτημα. Πού πάνε αυτά τα μικρά ψάρια, ξαϊλώνονται, χάνονται ή μήπως εξάγονται παράνομα. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αν όλοι ακολουθούσαν τους κανόνες δεν θα υπήρχε βέβαια πρόβλημα. Κύριε Νίλσον, σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας ε, και νομίζω ότι μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για το τι πρέπει να κάνουμε όσον αφορά την ε, λισαβονοποίηση ή όχι και στις προηγούμενες εκθέσεις είχαμε λισαβονοποίηση και μπήκαμε σε λεπτομέρειες και επιτύχαμε αλλαγή. Νομίζω ότι όλοι συμφώνησαν επ' αυτού, άρα δεν νομίζω ότι εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Πολύ καλά. Αν δεν υπάρχουν άλλα θέματα, θέλω να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 25 Φεβρουαρίου, το μεσημέρι. Σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, ανέφερα μία εβδομάδα παράταση, αλλά δεν είπα πια η ημερομηνία ακριβώς. 4 Μαρτίου, λοιπόν, για την παράνομη αλία. Λοιπόν, και εδώ 25 Φεβρουαρίου επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν άλλα θέματα. Λύτε συνεδρίαση, μέχρι αύριο στις 9. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους καθώς και τους διερμηνείς. Γεια σας.